Okay, good afternoon, colleagues. Seems a bit of a slow start. It's people traveling on Mondays. Καθυστερήσαμε λίγο να αρχίσουμε. Καλή σα, ε, καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι. Βέβαια είναι και Δευτέρα απόγευμα και υπάρχουν αεροπλάνα και Όμω λοιπά. 3 και 35 έχουμε προσκεκλημένο ομιλητή, οπότε να αρχίσουμε. Μπορούμε να δούμε το θέμα 1. Δεν βλέπω να έχετε κοινοποιήσει ε, παρατηρήσει για την ημερήσια διάταξη, αλλά θεωρώ ότι εγκρίνεται. Σα ευχαριστώ πολύ. Ανακοινώσει. Τώρα έχω ορισμένε ανακοινώσει. Και πρώτα, τούτη την εβδομάδα, το Κοινοβούλιο οργανώνει Εβδομάδα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ε, με την 30η ε, επέτειο. 70η εννοεί ο επέτειο τη ε, προκήρυξη των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Τώρα το Δεκέμβρη στο Στρασβούργο δεχόμαστε τους βραβευμένους με το βραβείο ε, Ζαχάροφ. Αλλά δυστυχώς ο φετινός βραβευμένος ε, είναι στις φυλακές και δεν θα μπορέσει να ε, προσέλθει. Όμως η 70η αυτή επέτειος και η κατάσταση που βρισκόμαστε σήμερα μας δείχνει ότι έχουμε πάρα πολύ δρόμο ακόμη να κάνουμε. Η Επιτροπή μας ασχολείται με τα θέματα αυτά και ζητεί οι άνθρωποι να διαβητούν σε αξιοπρέπεια. Και γι' αυτό μιλούμε και για του στόχου τη ε, βιώσιμη ανάπτυξη. Και η Εβδομάδα Ανθρώπινων Δικαιωμάτων για μα είναι πάρα πολύ σημαντική. Έχουμε ορισμένα θέματα στην ημερήσια διάταξή μα που εντάσσονται σε αυτήν την εβδομάδα. Σε λίγο θα αρχίσουμε με τα δύο πρώτα επί της ουσίας θέματα μας για το δικαίωμα στην τροφή πρώτα. Και αύριο θα έχουμε παρουσίαση από την Επιτροπή Εξωτερικών Θέσεων για δεσμευτική συνθήκη για ε, διεθνή συνεργασία για τα δικαιώματα, για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έχουμε όμως και δύο έξτρα συνεδριάσεις οι οποίες θα γίνουν την Τετάρτη το απόγευμα. Τετάρτη απόγευμα λοιπόν στις 3 έως τις 5 το απόγευμα. Όλα τα μέλη της Επιτροπής μας προσκαλούνται σε ανεπίσημη συνάντηση με το δίκτυο Voice μη κρατικών οργανώσεων που εργάζονται για ανθρωπιστική βοήθεια και θα εξετάσουμε ευκαιρίες και προκλήσεις της Ευρωπαϊκής Ανθρωπιστικής Βοήθειας. Πρόκειται για την αίθουσα ASP3E3 e την Τετάρτη το απόγευμα. Την ίδια ημέρα προβλέπεται κοινή συνάντηση με την Επιτροπή Γεωργίας και θα αναφέρουν σχετικά με την ε, αποστολή που έγινε στη Μαδρίτη για θέματα ε, Πείνα στον κόσμο και υποσυτισμού. Και θα συζητήσουμε και με τον Τόμ Άρνολτ, επικεφαλής της Task Force για την ε, Υπέθριο Αφρική. Και αυτό θα γίνει στην αίθουσα 1α02 του κτηρίου PHS από τι 5 και 4 έως τις 6.30 το απόγευμα. Πάλι την 4η το απόγευμα. Παρακαλώ οι συνεργάτε των ε, των ε, Ευρωβουλευτών και το προσωπικό των κοινοβουλευτικών ομάδων να τα σημειώσουν αυτά για να τα μεταφέρουν στους Ευρωβουλευτές. Επίσης, ένα ας πούμε λυπηρό γεγονός, ένα, μια λυπηρή είδηση. Ορισμένοι από εσάς θα ακούσατε ότι ε, ε, δεν είναι, είναι ευχάριστο γιατί ο Μπόγκταν έγινε δήμαρχος στην Κίντσε, στην Πολωνία και εγκαταλείπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν είναι εδώ, αλλά ούτε και η ομάδα του εκπροσωπείται είμαι βεβαία ότι μπορούμε να σημειώσουμε στα πρακτικά τις ευχαριστίες μου στον Bogdan Βέντα για όλα αυτά τα χρόνια συνεργασίας του και εργασίας του εδώ στην Επιτροπή μας ως ε, ε, συντονιστή του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Είναι και τα γενέθλιά του σήμερα. Άρα, αν θέλετε, μπορούμε να του χρόνια πολλά όταν θα έρθει. Είναι βέβαια πολύ ε, πολύ άσχολο. είναι και η τελευταία του ημέρα σήμερα στο Κοινοβούλιο και επομένω έχει να κάνει πολλά πράγματα. Είμαι βεβαία θα τον δούμε αργότερα. Παρακαλώ όμω να εγγραφούν στα πρακτικά οι ευχαριστίε μου και οι ευχαριστίε της Επιτροπής μας τον Μπόγκταν. Όταν θα έρθει μπορούμε να πούμε λίγα λόγια τότε. Και άλλη μια ανακοίνωση, αλλαγή αυτή τη φορά στην γραμματεία μα. Η Πέτρα Ολμάιστερ, α εδώ είναι η Πέτρα, εκεί κάθεται με τα κόκκινα μαλλιά, που εργάζεται μαζί μας εδώ 13 χρόνια και θα μετακινηθεί από 1η Δεκεμβρίου στη Γενική Διεύθυνση Προεδρίας με τον, την κυρία Κόκλαντ. Πέτρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαστε εδώ πάρα πολλά χρόνια περισσότερα από όλες και όλους μας. Παρακαλώ να ευχαριστήσουμε την Πέτρα. και είμαι βεβαία ότι θα σε βλέπουμε όταν θα πηγαίνουμε να πάρουμε τις ε, κάρτες πιοφορίας. Είμαι βεβαία ότι θα σας βλέπουμε σε τέτοιες ε, περιπτώσεις. Τώρα, να περάσουμε στο θέμα 3. Α, έχω και άλλη ανακοίνωση. Στις, την Τετάρτη το απόγευμα πάντοτε οργανώνω μια εκδήλωση για ανθρώπινα δικαιώματα με την ε, μη κυβερνητική οργάνωση Global Witness για αυτούς που αγωνίζονται υπέρ των ανθρώπινων δικαιωμάτων και το φυσικό περιβάλλον. Θα σας στείλω και σχετικό σημείωμα. Στις 6 ώρα το απόγευμα ε, θα είναι μια καταπληκτική ε, φωτογραφική έκθεση των δραστηριοτήτων ε, των ανθρώπων αυτών. Θα σας στείλω και σχετικές πληροφορίες σε όλους. Τώρα, το υπαριθμό 3, έγκριση των πρακτικών. Έχετε τα πρακτικά της 23ης, 24ης, 4ου, 11-12 6 29 38 και 24-9. Αν έχετε σχετικές παρατηρήσεις, σας παρακαλώ να τις γνωρίσετε στην γραμματεία. Οι δεμοί θα θεωρηθούν τα, τα πρακτικά αυτά εγκεκριμένα. Υπάρχουν 4 αποφάσεις και συστάσεις των συντονιστών της 9 Οκτωβρίου 2018. Πάλι, αν έχετε σχόλια, μέχρι τέλους της συνεδριάσεως στην γραμματεία. Αλλιώς θα θεωρηθούν, εγκεκριμένα. Το 5, τώρα ανακοινώσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Α, Κάρστεν, εσείς έχετε το λόγο, ορίστε. Έχετε κάποια ανακοίνωση. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δύο ε, ζητήματα ε, για ενημέρωση των αξιοτήμων μελών σας. Στις 26 Νοεμβρίου διεξάγεται Συμβούλιο Πρώτων για θέματα ανάπτυξης και θα συζητηθεί μεταξύ άλλων η Συμμαχία Ευρωπαϊκής Ένωση Αφρικής για βιώσιμες θέσει ανάπτυξης και επίσης για ICI, για ε, ορισμένες πτυχές, καθώς θα προβλέπεται και γεύμα για θέματα ισότητας φύλων. Άλλο θέμα που θέλω να σας αναφέρω είναι η επικείμενη δημοσίευση από το OECDAC της European Peer Review. Ξέρετε ότι κάθε 5 ή 6 χρόνια, ας το πούμε αλλιώ. ο DAC ε, επανεξετάζει γίνεται επανεξέταση μάλλον ε, ε, αξιολόγηση των μελών μεταξύ τους και κάθε 5-6 χρόνια αλλάζει η σειρά και τώρα είναι η δική μας σειρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο ECDAC πρόκειται να δημοσιεύσει τα απορίσματα της αξιολόγησης αυτής περί τα τέλη του μηνός. Και είμαι βέβαιος ότι θα ενδιαφέρει το Κοινοβούλιο να ενημερωθεί. Άρα το σημειώνω αυτό για να το λάβετε υπόψη σας στον προγραμματισμό σας. Ευχαριστώ Κάρστεν για αυτό το OECD Peer Review θα οργανώσουμε εμείς ή δυνατόν συνάντηση τον Ιανουάριο, γιατί το Δεκέμβριο ούτως ή άλλως έχουμε ε, δυσκολία να προβλέψουμε συνεδριάσεις τον Δεκέμβριο. Θα το βάλουμε λοιπόν στη μερίσια διάταξη του Ιανουαρίου. Κανονικά, ε, προηγούμενες φορές έχουμε λάβει πολλές ε, ενημερώσεις από την κυρία Μογκερίνη, από η FAC-DEV. Έχουμε γράψει όμως την Υπηρεσία Εξωτερικών Δράσεων και έχουμε παρακαλέσει η κυρία Μογκερίνη να είναι διαθέσιμη για ενημέρωση των ευρωβουλευτών, ίσως σε συνάντηση των συντονιστών, για να έχουμε ενημέρωση για αυτή την πολύ σημαντική συνάντηση του Συμβουλίου, σημαντική για την Επιτροπή μας. Ελπίζω να μπορέσουμε να το κάνουμε στο Στρασβούργο του Δεκεμβρίου, δύο η ώρα το μεσημέρι της Τετάρτης. Σας ευχαριστώ λοιπόν, αυτές ήταν οι ανακοινώσεις. Τώρα, υπαριθμόν 6 όπου νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα λάβει το λόγο. Νομίζω ότι ε, έτσι είναι. Θα έρθετε εδώ να καθίσετε. Ωραία. Λοιπόν, το θέμα 6 της ημερήσιας διάταξης. Η εφαρμογή της ευρωπαϊκής πολιτικής για τρόφιμα και διατροφή. Ασφάλεια τροφίμων και διατροφής. Η τρίτη έκθεση αναδιετία. Για τα επόμενα δύο θέματα, και αυτά σχετίζονται με το δικαίωμα στην διατροφή και πάντοτε μέσα στα πλαίσια τη εβδομάδας ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εγώ είδα στο BBC αυτή τη Σαββατοκύριακο, είδαμε πάλι εικόνες παιδιών που λιμοκτονούν στην Ιεμένη και όχι μόνο παιδιών αλλά γενικά ανθρώπων. Είναι πάρα πολύ καθαρό ότι τα τελευταία τρία χρόνια έχει πάλι σηκωθεί, έχει πάλι γευθεί το φάσμα της πείνας ανά όλο τον κόσμο και αυτό θα τα πείτε κι εσείς και ο ο συγκεκριμένος μας σε λίγα λεπτά από όσα ακούμε και βλέπουμε είναι καθαρό ότι όσοι ασχολούνται με αυτά πρέπει να κάνουν περισσότερα πράγματα για να επιτύχουν τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης και δυστυχώς η επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια που δίνεται ε, μειώνεται για τη διατροφή δηλαδή, Α, το, από το 8% έχει κατέβει στο 6% το 2016, από 8% το 2014. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε, διότι έχουμε δει τα ίδια και με τη χρηματοδότηση για την εκπαίδευση. Μειώνεται δηλαδή σε πολύ θεμελιώδη πράγματα. Πάμε υποτίθεται να επιτύχουμε τους ε, στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, αλλά στην πραγματικότητα ε, καταβαραχρώνονται οι χρηματοδοτήσεις. Έτσι λοιπόν πρώτα θα ακούσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ειδικότερα από τη Γενική Διεύθυνση ΔΕΦΚΟ, για την τρίτη τους αναδιατία έκθεση των χωρών μελών της Ένωσης και της ε, λαμβάνουν ε, που αναλαμβάνουν για ασφάλεια τροφίμων και διατροφής. Υπενθυμίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι χώρες μέλη έχουν υιοθετήσει σχετικό πλαίσιο για την ασφάλεια προμήθεια τροφίμων του 2010 και ότι υπάρχει και σχέδιο από το 2013 και κατόπιν αυτού η πρώτη αναδιετία έκθεση προόδου δημοσιεύθηκε το 2014 με τις σχετικές έξι προτεραιότητες που προβλέπει η πολιτική αυτή. Έχουμε και έκθεση, ναι την έχουμε την έκθεση, ορίστε σας τη δείχνω αυτή τη στιγμή. Έχει διανεμηθεί στα μέλη της Επιτροπής, παρακαλώ να γίνει, να διανεμηθεί τότε, αν δεν έχει διανεμηθεί ακόμη, ορισμένοι την έχουν. Βλέπω ότι οι προτεραιότητες είναι ανθεκτικότητα των μικρών εκμεταλλεύσεων, διακυβέρνηση, υποστήριξη της περιφερειακής γεωργίας, μηχανισμοί κοινωνικής προστασίας, διατροφή και ιδίω για ε, μητέρες, μικρά παιδιά και παιδιά, συντονισμός μεταξύ ε, δρόντων στην ανάπτυξη και στον ανθρωπιστικό τομέα και ανθεκτικότητα και ε, ασφάλεια για την διατροφή και την ε, για διατροφή και τα τρόφιμα. Θα δώσω το λόγο πρώτα στην ε, κυρία Μίτσι της Γενικής Διεύθυνση ΔΕΦΚΟ, στον κύριο Μίτσι, με συγχωρείτε πολύ, που έχει έρθει, μάλλον έχει δει και στην Ιεμένη και αλλού. Γνωρίζω ότι είχατε πάει και στην Ουγγάντα και ε, όταν πήγαμε και εμεί είχαμε μιλήσει με ανθρώπου εκεί που μα είπαν ότι η κακή διατροφή των παιδιών έχει δεινές επιπτώσεις και στην και στην διατροφή αλλά και στην εκπαίδευση αργότερα. Κυρία Μοντέση, ορίστε παρακαλώ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το, τη δυνατότητα να σας παρουσιάσω αυτή την τελευταία μας έκθεση για την πρόοδο των προσπαθειών μας να χρησιμοποιήσουμε την αναπτυξιακή συνεργασία για την προώθηση της επιστημιστικής ασφάλειας. Είναι, όπως είπατε, ε, μια έκθεση για την οποία έχετε μια περίληψη, έχει ήδη διανεμηθεί και βεβαίω υπάρχει και το ε, αναλυτικότερο σκέλος της έκθεσης με όλα τα στοιχεία. Ήδη αναφέρατε ποιο είναι το σημαντικό ζήτημα, ότι αυτή τη στιγμή διαπιστώνουμε ότι δεν βελτιώνεται η κατάσταση της επιστημιστικής ασφάλεια, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν εκατομμύρια άνθρωποι οι οποίοι ε, κινδυνεύουν από λοιμό σε ολόκληρο τον κόσμο ότι το 2017 διαπιστώνουμε, από το 2007 μάλλον διαπιστώνουμε ότι το θέμα αυτό θα πρέπει να συνεχίσει να μας αποσχολεί, ότι η κατάσταση έχει επιδεινωθεί, ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε να δούμε, να βλέπουμε πώς θα το αντιμετωπίζουμε και στο μέλλον και στο, στους μελλοντικού μας ε, προγραμματισμό. Θα επανέλθω τώρα στην ε, έκθεση. Σωστά α, περιγράψετε το πλαίσιο μέσα στο οποίο τη δημοσιοποιούμε πρόκειται για μια έκθεση που αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη, επομένω συντάσσεται από κοινού. Και δείχνει με αριθμητικά στοιχεία τις προσπάθειες που έγιναν για να επιτύχουμε τους κοινούς μας στόχους. Κοινοί στόχοι οι οποίοι καθορίστηκαν το 2010 με την πολιτική ε, για την επιστημιστική ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το ε, σχέδιο εφαρμογή τη του 2013. Αυτό είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο εργαζόμαστε. Πρόκειται για μια έκθεση την οποία προετοίμασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά με συνεργασία των αρμοδίων για την ε, περιφερειακή ανάπτυξη στα κράτη-μέλη. Γίνεται μια συνάντηση των εκπροσώπων της Επιτροπής με τους εκπροσώπους των κρατών μελών και την αξιοποίησαμε αυτή τη συνάντηση για την προετοιμασία. Τι καλύπτει αυτή η έκθεση. Θα έλεγα ότι είναι αναλυτική. Περιγράφει τις εξελίξεις στον τομέα της πολιτικής και σε παγκόσμιο επίπεδο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο τα τελευταία δύο χρόνια. Ε, την πρόοδο που έχει σημειωθεί στον τομέα της εκταμίευσης ε, ποσών, στην επίτευξη προτεραιοτήτων που είχαμε θέσει, προτεραιοτήτων πολιτικής, ορισμένες ε, περιπτώσεις ε, ε, όπου η παρέμβασή μας ήταν επιτυχής, όπως για παράδειγμα στο Λάος, όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση και 7 κράτη-μέλη και η Ελβετία ε, δημιούργησαν και ακολούθησαν ένα πρόγραμμα από το 2006 μέχρι το 2020 για την ε, επιστημιστική ασφάλεια. Άλλα στοιχεία τα οποία είναι πολύ σημαντικά είναι η επίπτωση της κλιματικής αλλαγής και επίσης η γεωργία, οι πρακτικές στη γεωργία με τρόπο που να βοηθούν την επιστημιστική ασφάλεια. Είναι σημαντικό να αναδεικνύουμε τη σχέση που υπάρχει μεταξύ της επιστημιστικής ασφάλειας αφενός και της κλιματικής αλλαγής και των πρακτικών στην γεωργία αφετέρου. Θα επανέλθω. να περιγράψω συνοπτικά τώρα ποια, ποιο πρόοδο σημειώθηκε. Πλευράς οικονομικής, λαμβάνοντα υπόψη τις διάφορες δεσμεύσει και από πλευράς Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από πλευράς κρατών μελών, μπορούμε να πούμε ότι έχουμε τηρήσει τις ε, υποσχέσεις μας. Τις δεσμεύσει δηλαδή που είχαμε αναλάβει να αξιοποιήσουμε οικονομικά εργαλεία που προορίζονται ακριβώς για αυτόν τον σκοπό. Συγκρίνουμε δηλαδή τα αριθμητικά στοιχεία αυτή τη έκθεσης με την προηγούμενη. Διαπιστώνουμε ότι η χρηματική ενίσχυση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη τη ε, για την επιστημιστική ασφάλεια έχει αυξηθεί κατά 4,2 δισεκατομμυρία ευρώ, δηλαδή αύξηση 14,7% σε σχέση με το 2014 και 26, 24% από το 2012. Επίσης προσπαθήσαμε να δώσουμε μεγαλύτερη ε, έμφαση, να δοθεί προτεραιότητα στην περιοχή της υποσαχάριας Αφρικής και αυτό μεταφράζεται σε, μια, σε ένα ποσοστό 53% του συνόλου της επιστημιστικής ασφάλειας που δόθηκε το 2016 για την περιοχή αυτή. Κατά κύριο λόγο η υποστήριξή μας εστιάστηκε στην βελτίωση της ανθεκτικότητας και των δυνατοτήτων των μικρών εκμεταλλεύσεων, γιατί θεωρούμε ότι αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Η έκθεση περιλαμβάνει και 10 συστάσεις. που βλέπετε αυτή τη στιγμή στην διαφάνεια. Θα σταθώ σε ορισμένε από αυτές. Η πρώτη, προφανώς, είναι να συνεχίσουμε να αναδεικνύουμε την σημασία που έχει η επιστημιστική ασφάλεια και ε, να αναγνωρίζουμε ότι πρέπει να συνεχίσει να προσπαθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη της να έχουν μια παρέμβαση για το θέμα αυτό στην παγκόσμια συζήτηση. επιπλέον σύσταση αφορά τη σημασία που έχει να έχουμε μια προσπάθεια από κοινού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της και του ΟΗΕ για να αντιμετωπίσουμε κρίσεις αλλά επίσης και να αντιμετωπίσουμε τις επιπτώσεις που έχει η κλιματική αλλαγή καθώς επίσης και οι πρακτικές στη γεωργία που θα πρέπει να ακολουθούνται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια, να δημιουργούνται θέσεις εργασίας κτλ. Η να φέρει ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε πιο γρήγορα στην συμφωνία επί συγκεκριμένων δικτών που θα μας επιτρέψουν, να παρακολουθούμε την πρόοδο. Αυτή τη στιγμή, σήμερα, αυτό είναι, είναι δύσκολο σε ορισμένους τομεί. Γνωρίζουμε με ακρίβεια πόσα χρήματα ε, ε, αξιοποιούμε για το τομέα αυτό. Μπορούμε επίσης να μετρήσουμε το τελικό αποτέλεσμα, δηλαδή σε παγκόσμιο επίπεδο πόσοι άνθρωποι ωφελήθηκαν από αυτά τα προγράμματα, αλλά είναι δύσκολο να παρακολουθήσει κανείς όλα τους τα αποτελέσματα και θα πρέπει να το βελτιώσουμε αυτό. Και άλλα σημαντικά θέματα να δείχνει η έκθεση. Ένα από αυτά είναι η σημασία που έχει να συνεχίσουμε να προγραμματίζουμε την παρέμβασή μας από κοινού. Ανέφερα ήδη την, καλή, ε, την επιτυχία που είχαμε στο Λάος, αλλά φαίνεται ότι έχει προστιθέμενη αξία να ε, γίνεται από κοινού ο προγραμματισμός μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, σε όσο το δυνατόν περισσότερες χώρες, αλλά επίσης και καθιστώντας αυτόν τον αποκοινού προγραμματισμό πιο γρήγορο. Με προγραμματισμό από κοινού πιθανώς σε πιο χαμηλό επίπεδο ανακλάδο. Θα πρέπει να ε, δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση και να αναδείξουμε τη σχέση που έχει η ανθρωπιστική βοήθεια, οι προσπάθειες μας για την ανάπτυξη και οι προσπάθειες μας για την ειρήνη. Συνεργαζόμαστε και με την ΕΚΟ στον τομέα αυτό. Όσο και να έχουμε προσπαθήσει αυτό δεν αρκεί, αρκεί επομένως θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε. Επίσης, Όπω σα έλεγα, θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή στην σχέση μεταξύ τη κλιματική αλλαγή και ε, των αλλαγών στη γεωργία ε, και να δούμε με ποιον τρόπο μπορούμε να προωθήσουμε την ανάπτυξη αυτών των περιοχών με έξυπνη καινοτομία. Πρέπει να υποστηρίξουμε τις, ε, την ύπεθρο σε αυτές τις περιοχές το δυνατόν καλύτερα. Κάτι ακόμα που αναφέρει η έκθεση δεν είναι καινούριο, αλλά διαπιστώνουμε για άλλη μια φορά ότι τη σημασία που έχει η ισότητα των δύο φύλων, ότι η δυνάμωση των γυναικών και η ισότητα των δύο φύλων οδηγούν σε αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών. Πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας. Και όπως σας έλεγα, θα πρέπει να εντείνουμε αυτές τις προσπάθειες στο πλαίσιο του επόμενου πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι αυτό το πλαίσιο θα μας δώσει τη δυνατότητα να έχουμε τους πόρους που χρειαζόμαστε για να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα της επιστημιστικής ασφάλειας και τις δυσμενείς εξελίξεις που ήδη αναφέρατε. Στο άμεσο μέλλον θα προσπαθήσουμε επίσης να βελτιώσουμε το πλαίσιο πολιτικής που έχουμε στα χέρια μας. έχει σημειωθεί πρόοδος, αλλά έχουμε και πολλέ νέε προκλήσει να αντιμετωπίσουμε, έχουμε μια εμπειρία που μπορούμε να αξιοποιήσουμε. Φαντάζομαι λοιπόν ότι την επόμενη χρονιά θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε ε, το πλαίσιο πολιτική με πρόταση τη επιτροπή προ το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. ότι μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορώ να σα διαβεβαιώσω ότι συνεχίζουμε να προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε την ανθρωπιστικέ καταστροφές, τις φυσικές καταστροφές, τον λοιμό σε ολόκληρο τον κόσμο. Έχουμε δημιουργήσει μηχανισμούς για άμεση παρέμβαση. Τι τελευταίες δεκαετίες αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση και στην πρόληψη, δηλαδή να καταστήσουμε τους τοπικούς πληθυσμούς περισσότερο ανθεκτικούς, να είναι περισσότερο σε θέση να αντιμετωπίσουν τέτοιες ε, κρίσεις ή καταστροφές. Και με αυτόν τον τρόπο πρέπει να συνεχίσουμε να προσπαθούμε, να επιμείνουμε Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν τις προσπάθειές μας. Είναι η κλιματική αλλαγή, είναι οι δημογραφικές μεταβολές, είναι η μετανάστευση παγκοσμίω. Και πρέπει για αυτόν τον λόγο να συνεχίσουμε να προσπαθούμε ακόμα περισσότερο. Και από την πλευρά μας ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιθυμούμε να συνεχίσουμε την καλή συνεργασία που έχουμε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έτσι ώστε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα. Σα ευχαριστώ για το ενδιαφέρον που δείξατε για την έκθεσή μα αυτή, την οποία σα μοιράσαμε και βεβαίω να απαντήσω και πιο συγκεκριμένα σε ερωτήσεις αν έχετε για τα στοιχεία που αναφέρει η έκθεση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Maria she's indicated first. I give you the floor. Η Μαρία Χόιμπουκ έχει το λόγο καταρχήν. Σας ευχαριστώ πολύ. Α, μια στιγμή. Ναι, να φορέσετε τα ακουστικά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παρουσίαση της εκθέσεως. Τονίσατε για άλλη μια φορά αυτή την διασύνδεση ανάμεσα στην γεωργία και το κλίμα. Όμως εδώ στις συστάσεις στην έκθεσή σας, στην υπαριθμόν 4, αναφέρεται μεν η αλλαγή του κλίματος, αλλά το μόνο άλλο που λέει είναι ότι χρειάζεται προσοχή από το θέμα αυτό δηλαδή από πλευράς Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης και κρατών μελών. Για άλλες συστάσεις ζητείτε πολύ εντονότερα, πολύ περισσότερα. Αυτό σημαίνει εκ του αντιθέτου ότι τα Υπουργεία Αναπτύξεως και οι διάφοροι οργανισμοί των ε, κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποδίδουν πολύ περιορισμένη σημασία στην αλλαγή του κλίματος και στις επιπτώσεις στη γεωργία και ότι γι' αυτό το λόγο στις ε, τομεακές συναντήσεις με τις ε, δικαιούχους χώρες δεν φαίνεται καν το θέμα αυτό να εμφανίζεται, να, να ε, απασχολεί. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλες ελλείψεις και στις χώρες μέλη μας και υπάρχουν και πολλοί οι οποίοι διατείνονται ότι δεν συμβαίνει καν η αλλαγή του κλίματος. Θα ήθελα λοιπόν να έχω μια τοποθέτηση εκ μέρους σας. Δεύτερο, ερώτηση προς το Συμβούλιο διότι εξ όσων γνωρίζω θα υπάρξουν συμπεράσματα του Συμβουλίου για την έκθεση πρόοδου και θα ήθελα να μου πείτε τι μπορούμε να αναμένουμε ως συμπεράσματα του Συμβουλίου. Πώς θα τοποθετηθούν δηλαδή τα κέντρα βάρους. Πώς θα διαμορφωθεί η συζήτηση αυτή στο Συμβούλιο. ενώ τη συζήτηση για το θέμα του κλίματος. Και εάν έχουν γίνει συζητήσεις και για την οικολογία της γεωργίας. Υπάρχουν μέθοδοι πολλά υποσχόμενες. Και στο κείμενο των συμπερασμάτων του Συμβουλίου θα ήθελα να περιληφθούν διότι θεωρώ πολύ χρήσιμες. Ευχαριστώ, η Πρόεδρος. Ας ε, δοθούν οι απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις, σε αυτή την ερώτηση. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος και από το Συμβούλιο. Μάλλον όχι. Άρα μπορείτε να απαντήσετε εσείς. Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω τώρα γαλλικά. Σας ευχαριστώ για αυτή την ε, παρέμβαση, το θέμα αυτό το οποίο είναι ύψης της σημασίας. Ήδη έχουμε παρουσιάσει την έκθεση στο Συμβούλιο και το Συμβούλιο θα προβάλλει συμπεράσματα κατά τα τέλη Νοεμβρίου. Αυτή είναι η πρόθεσή του. Επίσης, ζητήσαμε το Συμβούλιο για τις κλιματικές αλλαγές. Θα δούμε λοιπόν στην τελική έκδοση της έκθεσης κατά πόσο οι κλιματικές αλλαγές αντικατοπτρίζονται. Αλλά υπάρχει θέληση από το Συμβούλιο να δημιουργήσει αυτό το ε, σύνδεσμο τον άρρηκτο σύνδεσμο με τις κλιματικές αλλαγές. Είναι γεγονός ότι η έκθεση δεν μπαίνει σε λεπτομέρειες, αλλά σήμερα οι κλιματικές αλλαγές βρίσκονται υψηλά στην ατζέντα μας και εκεί θα παραμείνουν. Λαμβάνοντα υπόψη και τον μελλοντικό προγραμματισμό. Είναι μία προτεραιότητα λοιπόν του γενικότερου προγραμματισμού και θα υπάρχει αυτή η αιτιώδη συνάφεια μεταξύ γεωργίας και κλιματικών αλλαγών. Φυσικά τον αντίκτυπο τον βλέπουμε και στις χώρες εταίρους. Και παρά το γεγονός ότι δεν υπήρχε πολιτικός αντίκτυπος σε υψηλό επίπεδο, είδαμε ότι από τις χώρες Σαχέλ η από το κέρας του ελεφαντοστού, οι χώρες ανταποκρίνονται ως και βλέπουν την αιτιώδη συνάφεια μεταξύ διατροφής και κλιματικών αλλαγών. Είναι μια σημαντική δράση και φυσικά καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια σε επίπεδο πολιτικού διαλόγου ως προς τις κλιματικές αλλαγές και του, τη σύνδεση αυτής των κλιματικών αλλαγών και της γεωργίας. Φυσικά θα πρέπει να γίνει μεγαλύτερη προσπάθεια έτσι ώστε αυτή η διασύνδεση είναι ακόμα πιο έντονη. Αλλά υπάρχει εξέλιξη και με το διάλογο με τις χώρες εταίρους. Βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλη ε, πρόοδος από αυτές τις χώρες που βλέπουν αυτή τη διασύνδεση. Και εγώ έχω μία ερώτηση Φυσικά, το να υπάρχει διατροφική ασφάλεια υψηλά στην ατζέντα μας σημαίνει ότι όταν γίνεται προγραμματισμός που αντικατοπτρίζει αυτό το συσχετισμό θα πρέπει να δούμε κατά πόσο υπάρχει και συσχετισμός μείωσης της χρηματοδότησης. Δηλαδή οι χώρες ζητάνε χαμηλότερη χρηματοδότηση σε αυτή την περίπτωση. Θα μας ε, μιλήσει και ο Σαλ Γκέρενς και ο Έγγελς για τα νέα προγράμματα. Πώς είμαστε σίγουροι ότι υπάρχει αυτή η αντιστάθμιση στην επόμενη επταετία, δηλαδή στην επόμενη προγραμματική περίοδο. Όπως είπατε, στο προγραμματισμό θα το δούμε, αλλά μεταξύ των ε, προτεραιοτήτων αυτό το θέμα θα πρέπει να τονιστεί. Είναι σημαντικό, δεν αφορά όλες τις χώρες εταίρους, αλλά είναι μία βασική προτεραιότητα για τις χώρες που ανακύπτουν αυτά τα ζητήματα. Και φυσικά θα πρέπει να ε, ε, καλυφθεί και το θέμα των κλιματικών αλλαγών σε όλες τις χώρες. Τώρα γίνεται μία παγκόσμια δράση δημοσιονομικής φύσης, αλλά στην, ε, στον επόμενο προγραμματισμό αυτή θα είναι ε, μία από τις βασικές προτεραιότητες για όλες τις χώρες εταίρους. Υπάρχουν άλλοι συνάδελφοι που θα ήθελαν το λόγο επί του θέματος. Φαίνεται πως όχι. Περιμένουμε τον επόμενο μιλητή. Ο κύριος Μπίσλι έχει αργήσει γιατί ε, συνδέονται αυτά τα ζητήματα. Να δούμε λοιπόν πού βρίσκεται, γιατί έχουμε τον κύριο David Beasley από το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Διατροφής. Ε, να δούμε λοιπόν πού βρίσκεται. Okay, colleagues, I'm very pleased. Εντάξει λοιπόν κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, με μεγάλη μου χαρά καλωσορίζω τον David Beasley που είναι εκτελεστικός διευθυντής του World Food Program, του Παγκόσμιου Προγράμματος Τροφίμων. Ανέλαβε την, ε, ανέλαβε την ε, θέση του αυτή μόλις πέρσι και πριν από αυτό ήταν ε, κυβερνήτης της Νότιας Καρολίνας. Τον γνώρισα πριν από λίγους μήνες και μου εξήγησε πώς ε, κατάφερε εκεί οι άνθρωποι να συνεργαστούν και αυτό ίδιο συνεργάστηκε με διάφορους ε, ε, άλλους ηγέτες για να επιτύχει συμφιλίωση, ειρήνη και οικονομική πρόοδο. Επανήλθε μόλις από την Ιεμένη και του είπα ήδη ότι θα έχουμε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να γνωρίσουμε, να μάθουμε δηλαδή τι γίνεται στην Ιεμένη. Τα συζητήσαμε και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και διαπιστώσαμε ότι δεν μπορεί να περάσει καν η βοήθεια. Αντιλαμβανόμαστε ποια είναι τα μεγάλα πολιτικά εμπόδια εκεί. Είμαστε ιδιαίτερα γνώμονε για τη δουλειά που κάνετε. Όταν μπήκατε στο World Food Program, είχαμε τέσσερι αιστείε πείνα στον κόσμο. Νότιο Σουδάν, Βόρεια Νιγηρία, Ιεμένη και Σομαλία. Παραμένει η κατάσταση πάρα πολύ ε, ε, ανησυχητική στην Ιεμένη και στο Νότιο Σουδάν. Ωστόσο το ε, World Food Program έχει καταφέρει να επιστήσει την προσοχή των μεγάλων φορέων της διεθνούς κοινότητας στο μεγάλο πρόβλημα αυτό. Έχουμε, ακούσαμε και την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για, το, για την διατροφή και την ασφάλεια της διατροφής και τονίσαμε ότι η πείνα ξυπνά ξανά στον κόσμο. David, έχετε το λόγο. Ορίστε παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ χαίρομαι που σε ξαναβλέπω και μετά από λίγες ώρες ύπνου βέβαια αντιλαμβάνεστε και με όλες αυτές τις συγκρούσεις ανά τον κόσμο πέρασα μόνο λίγες ημέρες στην Ιεμένη αλλά και στη Συρία και στον Νίγηρα και στο Μαλί, στο Τσάντ και σε άλλα μέρη του κόσμου όταν ανέλαβα τον ρόλο μου τώρα πριν από 1,5 χρόνο, κάθε και σκέφτηκα μια στιγμή. Αντιμετωπίζουμε τη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση ανά τον κόσμο από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η NSA που είναι η μεγαλύτερη ε, δωρήτρια λέει ότι θα μειώσει, θα μειώσει την ε, ανθρωπιστική βοήθεια και μειώνουν και το μισθό. Πού πάω εγώ τώρα και αναλαμβάνω την ε, δραστηριότητα αυτή. Πολλοί όμω με εξήγησαν για ποιο λόγο είναι κρίσιμη η ανθρωπιστική βοήθεια και η ασφάλεια τροφίμων για την σταθερότητα σε όλο τον κόσμο. Και αν δεν αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα τη σταθερότητα διατροφή, δεν θα υπάρχει καμία πλέον ασφάλεια σε καμία χώρα του κόσμου. Έτσι, 1,5 χρόνο αργότερα, να με εδώ είμαι πάλι ακόμη. Ε, θα μιλήσουμε για την Ιεμένη και για τη Συρία και για τις επιπτώσεις της έλλειψης ασφάλειας διατροφής και τι σημαίνει για ολόκληρο τον κόσμο. Αλλά αν μου επιτρέπετε να σας δώσω μια ευρύτερη προοπτική από τότε δηλαδή που άρχισα να ασκώ τα καθήκοντά μου. Ήταν 777 εκατομμύρια άνθρωποι που πεινούσαν στον κόσμο κάθε μέρα. Ε. Τα τελευταία δύο χρόνια ο αριθμός αυτός αυξήθηκε και έφτασε στα 821 εκατομμύρια ανθρώπων. Οι άνθρωποι που είναι πραγματικά πολυμοκτονούν, μπορώ να το πω έτσι. Ο αριθμός αυτός από 80 εκατομμύρια προδιετίας έχει φτάσει στα 124 σήμερα εκατομμύρια. Και η πρώτη ερώτηση είναι γιατί αυτή η κορύφωση της πείνας. Πάμε σε λάθος κατεύθυνση. Ενώ είχε γίνει τόση μεγάλη πρόοδος στο παρελθόν, στα τελευταία 200 χρόνια και ιδίω στα, στα τελευταία 40 με 50 χρόνια είχε γίνει τόσο σημαντική πρόοδος για την αντιμετώπιση της φτώχειας, για την αντιμετώπιση της πείνας, για τη βελτίωση της ασφάλειας της διατροφής. Οι συγκρούσεις, οι ανθρώπινες συγκρούσεις είναι η βασική αιτία. Είτε μιλείτε για την Συρία ή για τους Ροχίνγκια που εκεί βρέθηκα πριν από δυόμιση εβδομάδες. Θα μιλήσω για Εμένη και Συρία, Σομαλία, Νίγηρα, Βόρειο-Ανατολική Νιγηρία, 19 χώρες όπου σημειώνονται βαρύτατες συγκρούσεις. Και βέβαια η άλλη κινητήρια δύναμη της πείνας είναι οι ακραίες μορφές του κλίματος. ιδίω στην Σαχέλ, όπου η Σαχάρα προχωρεί προς τα κάτω, προς τα νότια και ε, βλέπουμε την απερίμωση, βλέπουμε τις πλημμύρες, θα τα είδαμε αυτά και στη Συρία, θα σας τα πω σε λίγο. πολλά προβλήματα, αλλά έχουμε και λύσεις. Και για αυτά θα σας μιλήσω σήμερα. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να κάνουμε τα ίδια πράγματα. Και αυτό βλέπω, ξέρω και από την οπτική των Ηνωμένων Πολιτειών. Θέλω να πω για τη χρηματοδότηση, γιατί μιλήσαμε ε, γι' αυτό με την πρόεδρο σας, από τους κυρίαρχους λόγους για τους οποίους με έπεισαν να αναλάβω το ρόλο αυτό, οι φίλοι μου με έπεισαν ότι εγώ μόνος μπορούσα να πείσω τη νέα Αμερικανική κυβέρνηση ότι το World Food Program που είναι κάτι λιγότερο από 6 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο η χρηματοδότηση ήταν 1,9 δισεκατομμύρια δολάρια. Αν χάσουμε 1,9 δισεκατομμύρια δολάρια, αυτό θα είναι καταστροφή για το παγκόσμιο πρόγραμμα επισήτησμου. Μπόρεσα λοιπόν να παρουσιάσω τα επιχειρήματα αυτά, μπόρεσα να αλλάξω τη γνώμη του Λευκού Οικού που τώρα έχει ταχθεί υπέρ της ασφάλειας τροφίμων και παρόλο που η Ουάσιγκτον φαίνεται να καταπολεμεί τους πάντες και τα πάντα, όμως ωστόσο έχει ταχθεί υπέρ της ασφάλειας της διατροφής. Έχω λοιπόν από τους ρεπομπλέγανους και Δημοκράτες, οι Δημοκρατικούς, οι οποίοι συνεργάζονται ε, στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ και ένα είδο ειρήνη έχει συναυθεί μεταξύ αυτών των δύο συγκρόμενων πολιτικών δυνάμεων. Από την σκοπιά των ΗΠΑ ανήλθε η συγχρηματοδότηση από 9,9 δι σε 2,5 δι φέτος. Και φέτο αναμένουμε να πάει από τα 2,5 περίπου στα 3 δισεκατομμύρια δολάρια. Και το μήνυμα που λαμβάνω από τους φίλους μας ε, στο Λευκό Οίκο, αλλά και από τους επικεφαλείς των Δημοκρατικών και των Ρεπουμπλικανών να πει, μας, είπε, μας μου είπαν στους Ευρωπαίους συμμάχους μας ότι εμείς αυξάνουμε την βοήθεια, να αυξήσουν και αυτοί. Και μπορώ να πω τώρα στους Αμερικανούς φίλους μας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία αυξάνουν και αυτοί την βοήθεια. Διότι όλοι μαζί πρέπει να συνεργαστούμε όλοι, μαζί βρισκόμαστε στην ίδια βάρκα Καμιά φορά φτιάχνουμε σιλό, φτιάχνει το ανθρωπιστικό σιλό, μετά φτιάχνει το ε, σιλό τη βοήθεια. δεν λειτουργούν έτσι τα πράγματα. Αυτά λειτουργήσαν για κάποια 30-40 χρόνια. Αλλά δεν είναι τόσο απλό πλέον σήμερα. μια κατεβήγουσα κατάσταση που οφείλεται ας πούμε σε μια φυσική θεομηνία ή καταστροφή ή σε μια σύντομη σύγκρουση μπορεί να αντιμετωπιστεί ενδεχομένως σχετικά εύκολα με ανθρωπιστική βοήθεια ή αν έχεις μακροχρόνια ανάπτυξη, αλλά η ευρύτερη περιοχή του Σαχέλ, όταν πήγα και μίλησα στην διάσκεψη ασφαλείας του Μονάχου πριν από μερικούς μήνες με τον Καγκάμε και όλοι μιλούσαν για τη Σαχέλ. Και ο Καγκάμε και ο πρόεδρος του Σρουάντα είπε, μα δεν είναι πρόβλημα τη Σαχέλ είναι πρόβλημα τη ευρύτερη Σαχέλ και μάλιστα από τον Ατλαντικό μέχρι την Ερυθρά Θάλασσα. Ε, σε όλη αυτή την ε, απόσταση έχουμε εύθραυστες κυβερνήσεις, εύθραυστα περιβάλλοντα, φυσικό, πολιτικό και αν συνδυαστούν όλα αυτά και με το Ισλαμικό κράτος το οποίο εξώνεται σιγά σιγά από την Συρία που πάνε κυρίως στην ευρύτερη περιοχή της Σαχέλ χέρι-χέρι με το Μπόκο Χαράμ και με την Αλκάιντα και προσπαθούν να εκμεταλλευτούν αυτά τα εύθραυστα περιβάλλοντα για να μας αποσταθεροποιήσουν. Γιατί γίνεται αυτό, διότι θέλουν να διεισδύσουν μέχρι, μέσω της αναγκαστικής μετανάστευσης. Και τα είδα αυτά και στη Συρία. Και είπα και στη γαλλική τηλεόραση προμηνών αν νομίζετε ότι έχετε πρόβλημα με τη Συρία, που λίγο πολύ είναι, ε, είναι λίγο παραπάνω από 20 εκατομμύρια, λόγω αποσταθεροποίησης, λόγω συγκρούσεων, λόγω μικράς διείζησης του Άισις, περιμένετε να δείτε τι θα γίνει με το Σαχέλ, με 500 εκατομμύρια κόσμο εκεί, αν αυτοί αποσταθεροποιηθούν. Μπορούμε να δρούμε Όπω να αντιδρούμε δηλαδή, όπως στη σύγκρουση της Συρίας, αλλά θα είναι εκατονταπλάσια η προσπάθεια που θα απαιτηθεί. Αντί να αντιμετωπίσουμε έγκαιρα τα πράγματα στη ρίζα του όπως με την οικονομική αποσταθεροποίηση, θα μπορέσουμε να εξοικονομήσουμε και πολύ περισσότερα χρήματα εν τέλει. Πάνω από 90 εκατομμύρια κόσμο διατρέφουμε καθημερινά πολλά μαθαίνει κανείς στην προσπάθεια αυτή για το πώς σκέπτονται οι άνθρωποι και το πώς πράττουν. Βρισκόμαστε λοιπόν επί τόπου, κάνουμε διαρκώς έρευνες και ένα πράγμα που διαπιστώσαμε στη Συρία είναι πρώτο, για κάθε 1% αύξησης της πείνα είναι 2% αυτοί που μεταναστεύουν περισσότερο, η αύξηση μετανάστευση. Δύο, δεν έχει καμία σημασία αν φεύγουν οι άνθρωποι από τη Συρία, από τον Ήγηρα. Δεν θέλουν να φύγουν από τι πατρίδε του. Δεν θέλουν να εγκαταλείψουν τι αιστείε του. Αν όμω δεν έχουν τρόφιμα, αν δεν έχουν ασφάλεια, θα κάνουν ό,τι είναι αναγκαίο για να προστατεύσουν τι οικογένειέ του. Εμεί είδαμε ότι κάθε Σύρο πριν να φύγει από τη Συρία είχαν μετακινηθεί τρει και τέσσερι φορέ μέσα στη Συρία. Εγώ πήγα σε στατόπεδα προσφύγων στην Ιορδανία και μίλησα με μια γυναίκα εκεί πριν από λίγε εβδομάδε και μου είπε ότι μετακινήθηκε 10 φορές μαζί με τα παιδιά της μέσα, από, μέσα στη Συρία. Πήγε σε διάφορους συγγενείς, διότι δεν ήθελαν να φύγουν. Χιλιάδες χρόνια ζουν στη Συρία. Δεν ήθελαν να εγκαταλείψουν τη χώρα τους, τελικά αναγκάστηκαν. Και υποστηρίζουμε ανθρώπους στη Συρία και, και είτε, πρόκειται, είτε είναι η Συρία, είτε η Ιορδανία, ο Λίβανος, η Τουρκία ένας σύρος στη Συρία μας κοστίζει 5 σεντ το γεύμα. Διπλάσιο κόστος λόγω του πολέμου. Είναι σε εμπόλεμες ζώνες. Διαπιστώσαμε ή μάλλον υπολογίσαμε ότι το κόστος της λειτουργίας μας σε αιτήσια βάση είναι ένα δισεκατομμύριο δολάρια υψηλότερο λόγω της αυξημένη, το αυξημένου κόστους της εφοδιαστικής λόγω των πολεμικών σειράξεων. Ένα δισεκατομμύριο δολάρια. Όμω, ένα σύρο στη Συρία μας κοστίζει 50 λεπτά, 50 λεπτά το γεύμα του. Ο ίδιο σύρο, 50 ευρώ, αν είναι στην Ευρώπη. Και ο σύρο του σιαλό δεν θέλει ο καημένο να είναι εδώ. Θέλει να είναι σπίτι του στη Συρία. Ένας τρόπος για να αντιμετωπιστεί η δυναμική της Συρίας είναι και ο εξής. 4 εκατομμύρια μετρικοί τόνοι στάρι παράγονται στη Συρία ανά χρόνο. Λόγω του πολέμου αλλά και λόγω του κλίματος έχουν κατέβει στο 1,2 με 1,4 εκατομμύρια μετρικών τόνων Μπορούμε να συζητήσουμε τέλος πάντων πότε θα λήξει ο πόλεμος, θα γίνει μετά, υπάρχουν βέβαια και πολλά κινούμενα τμήματα, ε, έχουν γίνει πάρα στατικέ στατικές κινήσεις γύρω-γύρω. Ε, πέρασα και από τη Δαμασκό πριν από λίγες εβδομάδες, πέρασα και από την Κούντα Δεν μπορείτε να πιστέψετε τι καταστροφή. Βλέπετε εικόνες στην τηλεόραση και είναι φρικτά, λέτε, μάλλον πρόκειται για μια εμμονωμένη εικόνα. Δεν είναι όμως. Ολόκληρη η περιοχή είναι κατεστραμμένη δίνουμε γεύματα σε σχολεία, προσπαθούμε να φέρουμε τα παιδιά πάλι στα σχολεία. Εδώ όμως νομίζω η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Δύση γενικότερα, πρέπει να κάτσει να σκεφτεί. Πρέπει να δώσει ξανά ελπίδα στον Συριακό λαό, χωρίς να υποστηρίξει το καθεστώς. Εμείς προσπαθούμε να σχεδιάσουμε προγράμματα τα οποία θα προσφέρουν ασφάλεια διατροφής για τους μικρούς γεωργούς, ανεξαρτήτως του ποιος ασκεί την πολιτική εξουσία σε οποιαδήποτε χώρα. Πρέπει να βοηθήσουμε δηλαδή τα αθώα θύματα του πολέμου, ανεξάρτητα από την πολιτική δυναμική του ποιος ασκεί την εξουσία δίνοντας έτσι, προσφέροντας έτσι ασφάλεια διατροφή σε οποιοδήποτε δεδομένο περιβάλλον, είτε στη Συρία όπου διατρέφουμε 3 εκατομμύρια ανθρώπων. Με τη δική σας βοήθεια υποστηρίζουμε, εσείς μας δίνετε ένα δισεκατομμύριο δολάρια φέτος. Υποστηρίζουμε 3 εκατομμύρια ανθρώπους με αυτά τα χρήματα στην Τουρκία. Με cash-based transfer systems, δηλαδή με μετρητά. 2 δισεκατομμύρια δολάρια τον χρόνο. Είμαστε το μεγαλύτερο παγκόσμιο ανθρωπιστικό πρόγραμμα. Όχι μόνο για προσφορά αγαθών, αλλά και για μεταφορά κεφαλαίων, με την έννοια ότι προσπαθούμε πάντα το να χρησιμοποιήσουμε τον καλύτερο τρόπο για την αντιμετώπιση της κάθε μια ανάγκης. Μπορώ να εξηγήσω, για παράδειγμα, ότι στην Τουρκία έχουμε χρεωστικές κάρτες που πιστώνονται με χρήματα και μπορούν να αγοράσουν οι πρόσφυγες ας πούμε να νοικιάσουν ένα σπίτι, μπορούν να αγοράσουν ε, τρόφιμα ή μπορούν να πάνε στο γιατρό. Ας πάρουμε το Λίβανο. Στον Λίβανο υποστηρίζουμε μα πολύ κόσμο και ο Λίβανος είναι μια μικρή και ευάλωτη οικονομία. με εκατοντάδες χιλιάδες πρόσωπα που υποστηρίζουμε στο Λίβανο. Εάν πάμε στο Λίβανο, με τα χρήματα που μας δίνετε και εσείς και το Ηνωμένο Βασίλειο, οι Γερμανοί, οι Ηνωμένε Πολιτείε και προσφέραμε μόνο προϊόντα, αγαθά, θα κατέρει η οικονομία του Λιβάνου. Πώς μπορούμε λοιπόν να ελαχιστοποιήσουμε την επίπτωση της ύπαρξης ενός εκατομμυρίου προσφύγων στο Λίβανο. Φτιάξαμε ένα cash-based system. Έχουμε φτιάξει 500 καταστήματα μικρά καταστήματα από την κοιλάδα Πεκά, οπουδήποτε βρίσκονται πρόσφυγες και τώρα αυτές οι εκατοντάδες εκατομμύρια δολαρίων που ξοδεύουμε στο Λίβανο, τα χρήματα αυτά πηγαίνουν και τα ξοδεύουν στο κατάστημα το οποίο τα προμηθεύεται από τον τόπιο αγρότη. Και το άλλο, το ένα τρίτο προέρχεται από τη διεθνή κοινότητα με κανονικές ανταλλαγές. Με τον τρόπο αυτό δηλαδή υποστηρίζουμε και στηρίζουμε την τοπική οικονομία. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ενισχύσουμε την οικονομία αντιμετωπίζοντας όχι μόνο την ε, ασφάλεια διατροφής αλλά και τις ανάγκες των προσφύγων. Τώρα στην ευρύτερη περιοχή Σαχέλ τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Διότι πιστεύουμε ότι κάθε ανθρωπιστική προσπάθεια θα πρέπει να είναι και μια ευκαιρία ανάπτυξης. Βλέπετε, τι μπορούμε να κάνουμε Έχω ένα μικρό βίντεο να σας δείξω αν θέλετε που θα, νομίζω θα σας φανεί εξαιρετικά ενδιαφέρον. Ορίστε. Yeah, you gotta get a little sound there. We can start it again if there's no sound. Oh, you have to put the sound up. I'll forget that guy.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

Maybe David will keep speaking and then we'll get... Ας συνεχίσει ο David και μετά βλέπουμε. Το βίντεο αυτό δείχνει πώς παίρνουμε τα ανθρωπιστικά δολάρια και τα κάνουμε ευκαιρίες για ανάπτυξη. Θα δείτε στην οθόνη. Είμαστε αυτή στην Νίγηρα. Είναι η Σαχέλ. Η εικόνα αυτή δείχνει πραγματικά πώ είναι το τοπίο σε όλη αυτή την ευρύτερη περιοχή της Αφρικής. Δεν είναι καμιά μεμονωμένη περιοχή αυτή. Αν εξετάσετε τα τελευταία 10, 20, 30, 40 χρόνια, η διεθνή κοινότητα έχει προσφέρει ανθρωπιστική βοήθεια και δεν φαίνεται να υπάρχει φως στο βάθος του τούνελ. Μπορεί να συνεχίσετε για τα επόμενα 40-50 χρόνια. Εάν όμως δεν υπάρξει μια ε, αναπτυξιακή λύση μαζί με την ανθρωπιστική δεν πρόκειται να κάνουμε τίποτα. Και η περιοχή αυτή είναι πολύ περίπλοκη. Πιο περίπλοκη ακόμη διότι η Σαχάρα επεκτείνεται με ρυθμό ένα χιλιόμετρο τον χρόνο προς νότον. Και αυτό σημαίνει ότι οι βοσκοί, οι νομάδες πιέζουν τους γεωργούς καθώς κατεβαίνουν. Έρχεται τότε το Ισλαμικό κρότο, ε, κράτος συγγνώμη, και εκμεταλλεύεται την κατάσταση αυτή καθώς και την έλλειψη νερού, την έλλειψη ευκαιριών αναπτύσσουμε μια τεχνική που λέγεται η μισέλινος. Είναι εντυπωσιακή, θα δείτε, διότι με το μέγεθος του World Food Program και στις περιοχές αυτές όπου διατρέφουμε εκατομμύρια ανθρώπους, ποτέ σχεδόν δεν βλέπω είτε σε refugee operation ή σε non-refugee operation, σε μια χώρα απλώς που είναι πάρα πολύ φτωχή, δεν θέλουν ε, ελεημοσύνες, θέλουν την ελευθερία τους, θέλουν, θέλουν βιωσιμότητα, θέλουν ανεξαρτησία. Όταν ερχόμαστε λοιπόν να προ, προωθήσουμε ένα πρόγραμμα Food for Asset, είτε με ευρώ είτε με δολάρια, δεν ενδιαφέρονται για την διαφορά αυτή. Θέλουν ελευθερία και ανεξαρτησία, θέλουν μια λύση. Η ανθρωπιστική βοήθεια και μόνη σε αυτά τα περιβάλλοντα που δεν είναι short term, δεν είναι βραχυπρόθεσμα, δεν αρκεί. Χρειάζεται μια μακροπρόθεσμη δυναμική. Σε αυτού του είδους τις περιοχές που του ξαναλέω η Μισελίνο έχει το σήμα της Μισελίνου όπως θα δείτε όταν ερχόμαστε με το πρόγραμμα αυτό Food for Asset θα δείτε τι γίνεται εάν το βάλετε μαζί με το πρόγραμμα διατροφή στα σχολεία είναι πραγματικά εντυπωσιακέ οι συνέπειε. Ε, μαθηματικά μπορούμε να το αναλύσουμε και να σα δείξουμε τι τρομερέ εξοικονομήσει. Ιδού τι θα ξοδέψετε για μια εικοσαετία. Αν προχωρήσετε όμω σε ένα οικονομικά αποτελεσματικό πρόγραμμα, μπορείτε να μιλάτε για efficiency όσο θέλετε. Μπορείτε να είσαστε 100% efficient, αλλά με μηδενικά αποτελέσματα. Ενώ αυτό που συζητούμε εδώ είναι πραγματικά αποτελεσματικά, αποδοτικά προγράμματα. Εγώ θέλω το World Food Program να φύγει από την business. Θέλω να υπάρχει στρατηγική, αναπτυξιακή στρατηγική για να φτάσουμε σε μηδενική πείνα. Ποια είναι η στρατηγική εξόδου, exit strategy. Με αυτά τα project της ημισελήνου, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Πέρσι διότι πρέπει να ενισχυθεί η πλευρά της ανάπτυξης από, περισσότερο από την ανθρωπιστική. Χρειαζόμαστε και τις δύο. Αλλά πρέπει να υπερισχύσει η αναπτυξιακή. Μιλήσαμε για αναδάσωση. Μόλις φυτέψαμε το δισεκατομμυριστό δέντρο. Έχουμε αποκαταστήσει πάνω από μισό εκατομμύριο εκτάρια γης χιλιάδες επί χιλιάδων εκταρίων γης. Τα έχουμε ξανακαταστήσει εκμεταλλεύσιμα. Φτιάχνουμε σημεία ίδρευσης, φτιάχνουμε δρόμους για να μπορούν να μετακινηθούν τα προϊόντα. Με τα δικά σας χρήματα, με τα χρήματα των δωρητών από τις ΗΠΑ. Δημιουργήσαμε 17.000 χιλιόμετρα οδών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά ε, εμπορευμάτων και ε, τροφίμων. Για αρδεύσεις, για διάβλους, για κανάλια δηλαδή αρδευτικά. Όταν ερχόμαστε λοιπόν με τα αποτελεσματικά αυτά προγράμματα Food for Asset φροντίζουμε να πάνε και τα παιδιά στο σχολείο. Εάν δεν υπάρχουν σχολεία, τα κορίτσια δεν έχουν καμία πιθανότητα να επιτύχουν. Να επιτύχουν. και κοριτσάκια λοιπόν τότε πάνε στο σχολείο και έρχονται αγορά και κοριτσάκια από διαφορετικέ φυλέ όπου κάθονται και τρώνε μαζί και έρχονται επομένω πολύ πιο κοντά. Όταν έχουμε λοιπόν τέτοια αποδοτικά προγράμματα, γνωρίζουμε και μα το δείχνει η εμπειρία, τότε η μετανάστευση εξαφανίζεται από του από τους χάρτες. Οι εγκυμοσύνες των πολύ νεαρών κοριτσιών, η αναγκαστική γάμοι των 12χρονων κοριτσιών εξαφανίζονται. Συγκρούσεις μεταξύ ε, αγροτών και κτηνοτρόφων μειώνονται, διότι επιλέγουμε πρώτα εκείνες τις περιοχές όπου μπορούμε να βοηθήσουμε να συνεργαστούν κτηνοτρόφοι με ε, γεωργούς. Ο Άισις εξαφανίζεται. Έχω περισσότερες μανάδες που μου λένε «Κύριε Μπίσλη, ο σύζυγός μου δεν ήθελε να πάει στο Ισλαμικό κράτος, στον Άισις, αλλά έπρεπε να ταΐσουμε το μωρό». Δεν ήξερε ο άντρας μου τι άλλο να κάνει. Όταν βρισκόμαστε λοιπόν εκεί, είμαστε η πρώτη γραμμή άμυνας κατά του εξτρεμισμού. Πιστεύω λοιπόν ότι αν μπορούμε να συνεργαστούμε σε συνεργασία και να συνεκάνουμε να συνεργαστούν ο ανθρωπιστικός με τον αναπτυσιακό τομέα, να μειωθεί η αναγκαστική μετανάστευση και να περιοριστεί στη μετανάστευση που γίνεται ε, με τη θέληση του ατόμου. Και αυτό τότε θα είναι μια πολύ πιο ευχάριστη συζήτηση. Είτε πρόκειται για την Κεντρική Αμερική, είτε πρόκειται για τις υπήρου σα. Μπορούμε ίσως να δούμε το, το βίντεο. Α, φαίνεται πως μπορούμε να το δούμε τώρα. Ωραία. Oh yeah.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 That two minute video, the visual. Σε αυτά τα δύο λεπτά είδατε πολύ ξεκάθαρα τη διαφορά ανάμεσα στο πριν και το μετά. Conflicts, riots, not me. terrorist attack. It's gone. Yeah. So, but the point of that video. Λοιπόν, αυτό που δείχνει αυτό το είναι ότι το Παγκόσμιο Επιστηστικό Πρόγραμμα έχει τη δυνατότητα, τις δυνατότητες να εφαρμόσει τέτοιου τύπου προγράμματα σε ολόκληρες περιοχές, μεγάλες περιοχές του κόσμου. Και αν αυτό συμβεί αποτελεσματικά, ε, είναι και πολύ οικονομικότερο σε σχέση με αυτό που κάναμε στο παρελθόν. Μπορούμε να εξοικονομήσουμε μακροπρόθεσμα πολλά χρήματα. Αυτό εννοώ όταν λέω ότι δεν πρέπει να υπάρχει πλέον απομόνωση μεταξύ της παρέμβασης της ανθρωπιστικής και της παρέμβασης για την αναπτυξιακή συνεργασία. Ε, την ίδια συζήτηση έχουμε και στις Ηνωμένε Πολιτείε για το πώς θα πάψουν να υπάρχουν αυτά τα σιλό, αυτή η διάσπαση των δυνάμεών μας, γιατί δεν βρισκόμαστε πια στην ίδια κατάσταση όπως βρισκόμασταν πριν 50 χρόνια. Χρειάζεται κανείς μακροπρόθεσμα να έχει ευέλικτο τρόπους να δημιουργήσει μακροπρόθεσμες λύσεις. Να σας δώσω και λίγες πληροφορίες για την Ιεμένη. Βρισκόμουν εκεί πρόσφατα. Ε, και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ που συζητά την κρίση την ανθρωπιστική στην περιοχή, η οποία επιδεινώνεται παρά το γεγονό ότι το επίπεδο των συγκρίσεων παραμένει το ίδιο, έχει αλλάξει η δυναμική. Ε, η, η Εμένη ήταν μια φτωχή χώρα εδώ και πάρα πολύ καιρό, πολλά χρόνια. Ε, υπήρχαν δηλαδή πολύ σημαντικά προβλήματα φτώχεια ακόμα και πριν ξεκινήσει ο πόλεμος. Βρισκόταν πολύ ψηλά στο, στις, στις χώρες με τέτοιου τύπου προβλήματα και να γλαγματίσω ότι μία του Ριάντα έχει κατακριμνιστεί από ένα δολάριο που αντικατοικούσε σε 11 ε, τώρα έχουν φτάσει στο ένα δολάριο να αντιστοιχεί στα 250. Ε, στην αρχή του, πολέμου αυτό και τώρα στα 720. Έχει επηρεαστεί σύγκρουση σε μεγάλο βαθμό από την πολιτική της Σαουδικής Αραβίας, η οποία έχει επιβάλλει αποκλεισμό και δεν παρήχε οικονομική βοήθεια. Αυτή τη στιγμή έχουμε τα χρήματα που χρειαζόμαστε, όμως δεν μπορούμε να τα να ε, παρέμβουμε στο πεδίο. Γιατί υπάρχουν περιοχές στις οποίες δεν μπορεί κανείς να ε, έχει πρόσβαση ανάλογα με το με ποιον συνεργάζεται. Ποιο είναι το πρόβλημά μας λοιπόν τους τελευταίους μήνες ο αριθμός που κινδυνεύει με λοιμό ε, αυξάνεται δραματικά. Τους τελευταίους τρεις μήνες αυξήθηκε αυτός ο αριθμός κατά 3,6 εκατομμύρια. 1,3 εκατομμύρια τις τελευταίες ημέρες. Ή 1,6 δεν είμαι σίγουρος. Αλλά ε, ε, είναι δραματική η αλλαγή. Μιλούμε για ανθρώπους που βρίσκονται στα όρια του λοιμού. Από 8 εκατομμύρια που είχαμε και υποστηρίζαμε, έχουμε φτάσει πλέον σε περίπου 12 εκατομμύρια ανθρώπους στα όρια του λοιμού. Και πεθαίνει τουλάχιστον ένα παιδί κάθε 12 λεπτά. Η κατάσταση είναι φιαλτική. Το δίλημα που αντιμετωπίζουμε είναι το εξή. Φαίνεται ότι δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τι ανθρωπιστικέ ανάγκε του πληθυσμού μόνο με ανθρωπιστική βοήθεια. Θα χρειαζόμαστε 100 με 150 εκατομμύρια δολάρια μόνο, μόνο για να αντιμετωπίσουμε τι ανάγκε των 12 εκατομμυρίων ε, ε, πολιτών τη Ιεμένη που λιμοκτονών. Οι συζητήσει που είχαμε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ήταν ε, θετικέ. Προσπαθούμε να βρούμε τρόπους να συνεργαστούμε για να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί και να βοηθήσουν και αυτή, αυτό ήταν πολύ θετικό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ηνωμένε Πολιτείε, ιδιαίτερα το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία ή η Ιαπωνία έχει συνεισφέρει, η Σαουδική Αραβία έχει επίσης ε, συνεισφέρει, όμως θα φτάσουμε τα 150 εκατομμύρια που χρειαζόμαστε ανά μήνα Ένα ποσό το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για αναπτυξιακή βοήθεια ανά τον κόσμο. Η ανησυχία μου όμω είναι η εξή, ότι εξαιτία τη ανθρωπιστική καταστροφή έχουμε και κατακριμνισμό τη οικονομία. Σα μίλησα για τη αναγνωματική ισονοτιμία. Αντίστοιχα προβλήματα έχουμε με την αγοραστική ε, δύναμη των πολιτών. Έχουν, έχουν χάσει οι πολίτε το 2 τρίτα τη αγοριστική του ισχύω. και μπορεί εμείς να καλύπτουμε 12 εκατομμύρια, αλλά 21 εκατομμύρια πρέπει να αγοράζουν τα τρόφιμά τους, ε, ενώ η ανεργία αυξάνεται με δραματικούς ρυθμούς. Και στον ιδιωτικό τομέα και αντίστοιχα προβλήματα υπάρχουν για όλους τους πολίτες. Η βοήθεια, κάποια μικρή βοήθεια ε, υπόσχονται τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και η Σαουδική Αραβία. Δεν υπάρχει λύση σε αυτό το πρόβλημα εάν δεν βρούμε κάποιο τρόπο να αυξηθεί η ρευστότητα στην οικονομία. Οι οικονομολόγοι μελέτησαν την περίπτωση τη Σιμένη και εξήγησαν στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ότι δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπίσουμε την ανθρωπιστική καταστροφή μόνο με ανθρωπιστική βοήθεια. Αυτή τη στιγμή χρειάζεται, φαίνεται, σχεδόν 200 εκατομμύρια δολάρια το μήνα να, ρευστότητας να εισάγονται στην οικονομία της χώρας έτσι ώστε να ε, επανέλθει η συναλλαγματική ισοτιμία και να σταθεροποιηθεί στο 1 δολάριο προς τα 300-450 έτσι ώστε να σταθεροποιηθεί η οικονομία και να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε cash-based ε, transfers όπως Σα περιέγραφα πριν. Και προσπαθούμε να δούμε πώς μπορούμε να συνεργαστούμε με τον Ηνωμένα Αραβικά Μιράτα, με άλλους δωρητέ για να το επιτύχουμε. Έχετε δει και με τα μάτια σας τις φρικτές εικόνες των παιδιών, τι εμπόλεμες ζώνες, τις πόλεις φαντάσματα. Δεν είναι, σας, μας θυμίζουν τις πόλεις φαντάσματα που βλέπει κανείς σε κινηματογραφικές ταινίες, σε western. η προσπάθεια Χούτι να βρουν καταφύγιο σε αποθήκες επειδή γνωρίζουν ότι τουλάχιστον εκεί δεν θα τους επιτεθεί κανείς να προστατευτούν από ελεύθερους κοπευτές. Εχτες και μόνο βρήκαμε επτά νάρκες τις αποθήκες που είχαμε για τα σιτηρά για την περιοχή που καλύπτει θεωρητικά ολόκληρη την περιοχή αυτούς τους 8 ε, εκατομμύρια ανθρώπους, 7 ανάρκες κατά προσωπικού σε περιοχή την οποία ελέγχουν οι Χούτι και στην οποία γνωρίζουμε ότι χρησιμοποιούνται νάρκες. Πώς γίνεται αυτό. Είναι απαράδεκτο. Βλέπω παιδιά σε νοσοκομεία, σε ένα θάλαμο, είδα ένα παιδί που είχε βάρος 3,3 κιλά, ενώ κανονικά θα έπρεπε να είναι περίπου 19 κιλά. Προσπάθησα λίγο να τον κάνω να χαρεί, να, χαμογελάσει. Ήταν σαν να μιλούσε σαν ένα φάντασμα. Δεν, δεν, δεν είχε ζωή αυτό το παιδί. Και αυτό που άκουγα από όλες τις Μητέρε από όλους τους σου εκεί είναι φροντίστε να σταματήσει ο πόλεμο. μη φύγετε. Και ρώτησε γιατί να μην φύγω. Ε, γιατί όσο βρίσκεστε εσείς εδώ, εξασφαλίζεται η ειρήνη. Και φροντίζουν να παίρνουν από εμάς το φαγητό ενός ολοκλήρου μήνα, γιατί είναι επικίνδυνο να έρχονται στις εγκαταστάσεις μας πιο συχνά. να προσπαθήσαμε να υποφεληθούμε τους παρουσίας μου εκεί που εξασφάλιζε μια κάποια ασφάλεια. Γιατί διαφορετικά και οι ίδιες οι δυνάμεις του ΟΗΕ τους αποθαρρύνουν. Μην πηγαίνετε στις ε, εγκαταστάσεις εκεί, είναι επικίνδυνο πολύ. Την άποψή μου πρέπει να το ακούσει ολόκληρο ο πλανήτης. Πρέπει να προστατεύσουμε αυτούς τους ανθρώπους οτιδήποτε και αν κοστίζει. Βεβαίω υπάρχουν διαφορέ μεταξύ των ομάδων των αντιμετωχόμενων, των Χούτι. Υπάρχουν ορισμένε με τι οποίε έχουμε μια αποτελεσματική συνεργασία για να περνάει ανθρωπιστική βοήθεια, αλλά υπάρχουν και άλλε τι οποίε ειλικρινά πρέπει να σα πω ότι να αν, αν, του ενδιαφέρει οτιδήποτε άλλο. Ε, έτσι έχουν τα πράγματα στο πεδίο στην Ιεμένη. Στα 3,5 χρόνια του πολέμου, ε, αυτό που δεν συνέβη μάλλον, με τα 3,5 χρόνια του πολέμου στην Ιεμένη θα συμβεί του επόμενου μήνε εξαιτία τη κατάρρευση τη οικονομία σε συνδυασμό με την ανθρωπιστική κρίση. Επομένω, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό και στο επίπεδο της οικονομία και στο επίπεδο τη ανθρωπιστική βοήθεια. Σα ευχαριστώ που μου δώσατε τη δυνατότητα να μιλήσω λίγο περισσότερο και να σα ενημερώσω για την κατάσταση με τι συγκρούσει ανά τον κόσμο, για το πόσο σημαντικό είναι να συνδυάσουμε την αναπτυξιακή βοήθεια με την ανθρωπιστική παρέμβαση, πόσο σημαντική είναι η παρέμβαση τη Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτή την προσπάθεια και σα ε, ευχαριστούμε για την ε, βοήθεια που δίνετε στο πρόγραμμα δικό μα και θα πρέπει να δούμε πώ μπορούμε να συνεργαστούμε καλύτερα. Επίση πρέπει να σα πω ότι το Παγκόσμιο Επιστημιστικό Πρόγραμμα θεωρείται ε, το καλύτερο από πλευράς διαφάνειας μεταξύ 500 διακυβερνητικών οργανισμών σε ολόκληρο τον κόσμο. Σας ευχαριστώ. Well, thank ευχαριστούμε πολύ. David, μας έδωσες όχι μόνο γνώση για την κατάσταση, την επιτόπια κατάσταση, αλλά κατέστησε σαφές ότι τα πρέπει να σταματήσουν. Πρέπει να έχουμε μια ολιστική προσέγγιση. Όχι να βλέπουμε μέρη του παζλ, Ευρωπαϊκή Ένωση, ΙΠΑ, Αφρική και ούτω καθεξής. Πρέπει να υπάρχει ολιστική προσέγγιση. Έχουμε δύο διευθυντές εδώ από την DG ECO και από την Γενική Διεύθυνση DEVCO που εργάζονται ως προς αυτούς τους, αυτή τη, σύνδεση όλων των πτυχών. Είδαμε λοιπόν πώς έχει η επιτόπια κατάσταση, είδα τι κάνατε και στην Τουρκία, στα σύνορα με την Συρία και φυσικά είναι πολύ πιο αξιοπρεπές να δώσει κανεί στου ανθρώπους χρεωστικέ κάρτες για να μπορέσουν να αγοράζουν το φαγητό τους και να ζήσουν όπως θέλουν. Αυτές οι ταμιακές μεταφορές ε, έχουν καταδικαστεί από πολλούς, αλλά θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι αυτό έχει καλύτερη επίπτωση σε ολόκληρη την οικονομία και φυσικά οι άνθρωποι που θέλουν ε, να παραμείνουν να μπορέσουν να μείνουν στη χώρα τους με αυτές τις κάρτες και η εργασία σας είναι μέρος αυτού του στοιχήματος. Ελπίζω να έχετε χρόνο να παραμείνετε για τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις. Η, Μίρια ε, Μύρια Βίκα Πέιβερ, ο κύριος Γκέρνενς, ο κύριος Πέτερλε, γιατί έχουμε μείνει πίσω. Αλλά και η κυρία Σόφκο, βεβαίως. Θα μιλήσω φινλανδικά, αν ε, μπορώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ για αυτή την ε, παρουσίαση ειλικρινή δίκαιη, αντικειμενική όσον αφορά τον λοιμό. Είπατε ότι πρόκειται για μάστιγα που προκαλεί ο άνθρωπος, ο πόλεμος, η πόλεμη, η ανθρωπιστική κρίση, η κρίση διατροφής, το θέμα της ξηρασίας και οι δυσχερείς καταστάσεις στην Αφρική όπου έχουμε και εσωτερική μετανάστευση, αλλά ε, πολλές είναι οι ρίζες της ε, κακοδαιμονίας. Για αυτή την ιδιαίτερα λυπηρή κατάσταση μας δώσατε στοιχεία τα οποία τρομάζουν. Ο λοιμός, το φάσμα της πίνας διωγγώνονται συνεχώς. Ως προς το πλαίσιο των λύσεων. Ήδη έχουμε φτάσει στο φεγγάρι, έχουμε ε, διάφορα προγράμματα, δορυφορικά προγράμματα, προγράμματα σε άλλους πλανήτες, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο η τεχνολογία θα μπορούσε να μας δώσει λύσεις που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε και σε περιοχές που γνωρίζουν την απερίμωση αυτή τη τεχνολογία τη γνωρίζετε στην ε, Αμερική και στην Ευρώπη. Ασχολούμαστε με την ε, τεχνητή νοημοσύνη, όπως την περίπτωση οχημάτων χωρίς οδηγό και ούτω καθεξής. Αλλά νομίζω ότι η τεχνολογία θα πρέπει να μας βοηθήσει για την εξάλληψη της πείνας θα μπορούσαμε να σκεφτούμε την αναδάσωση αυτών των περιοχών, για παράδειγμα, με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Επίσης, έχει μεγάλη σημασία η στοχοθέτηση αυτής της βοήθειας, έτσι ώστε αυτοί που λιμοκτονούν να λαμβάνουν την ε, βοήθεια αυτή. Δηλαδή υπάρχουν τρόφιμα σε παγκόσμια κλίμακα, αλλά δεν φτάνουν σε αυτούς που πρέπει να φτάσουν. Γι' αυτό πρέπει να γίνει στοχοθέτηση και να μπορέσουμε να δούμε επιτόπια πώς θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους πληθυσμούς που χρειάζονται πολύ περισσότερο την επισητιστική βοήθεια. Ευχαριστούμε πολύ Μαρία Χόιμπουκ ευχαριστώ πολύ. Σας γνωρίζω, γνωριζόμαστε κύριε ε, Διευθυντά, έχετε έρθει και στο γραφείο μου. Είναι πραγματικά ε, φρικτά τα σενάρια αυτά που μας δείξατε. Τώρα, όταν πηγαίνετε ως παγκόσμιο πρόγραμμα τροφίμων, ε, δεν περίμενα και τίποτε λιγότερο, ή αυτά που κάνετε είναι σωστά. Περίμενα ωστόσο να διευρύνετε την έκθεσή σας, δηλαδή να διασυνδέσετε περισσότερο την ανθρωπιστική βοήθεια με τα ε, αναπτυξιακά προγράμματα. Δείξατε και το βίντεο το οποίο το βλέπω εγώ για δεύτερη φορά, πολύ ενδιαφέρον, όπου δίνεται όντως υποστήριξη ε, στους αγρότες και τις αγρότησες. η καλύτερη οργάνωση θα είναι πραγματικά να μπορούν να καλλιεργήσουν τη γη τους τόπου. Οι ερωτήσεις μου είναι οι εξή. Ποιο ρόλο παίζει η βιοπικιλότητα στην εργασία σας, διότι είναι κύριο θέμα όταν μιλούμε για παραγωγή τροφίμων. Δεύτερο, μας δείχνετε στην ταινία πως καθοδηγείτε τους ανθρώπους ε, να ε, καλλιεργήσουν ε, την υγεία τους ε, με τι σπόρα, με τι σπόρους δηλαδή κάνουν την καλλιέργεια αυτή. Είναι σπόροι από ντόπιε παραγωγές. Τι είδου εκπαίδευση γίνεται για τις αγρότες και τους αγρότες. Υποθέτω ότι είναι ε, προσαρμοσμένοι στις ανάγκες. Και τέλος θα ήθελα να γνωρίζω με ποιες ιδιωτικές επιχειρήσεις συνεργάζεστε. Είναι οι τοπικές, είναι οι πολύ μεγάλοι διεθνείς όμιλοι οι οποίοι διαθέτουν κάποια πράγματα από εδώ και από εκεί πώς διαμορφώνονται οι λεπτομέρειες, διότι εδώ βλέπω εγώ να υπάρχει ένα σημαντικό, μια σημαντική δυνατότητα μόχλευσης για την, ανθρωπι... για την αναπτυξιακή βοήθεια. Σαλ Γκέρενς. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Μετά από αυτή την ε, μαρτυρία που μας συγκίνησε, θα πρέπει να έχουμε μία προσέγγιση κρατώντας αποστάσεις για να τονίσουμε και τις ρίζες του κακού. Εδώ και δέκα χρόνια είχα, ήμουν επικεφαλής του κλαμπ του Σαχέλ και είχαμε κάνει μία ε, έρευνα, δηλαδή τις τρεις δεκαετίες 60-90 ως προς τη γεωργική παραγωγή. Είδαμε λοιπόν ότι υπήρχε στασιμότητα. Η γεωργική παραγωγή είχε παραμείνει ίδια κατά κεφαλή. Αυτό ήταν ένα συμπέρασμα εκ πρώτης όψεως, αλλά είδαμε παράλληλα ότι είχε τριπλασιαστεί ο πληθυσμός. Άρα η γεωργική παραγωγή ήταν επιτρία σε σχέση με τις τρεις αυτές δεκαετίες. Μιλήσατε για το δημογραφικό, αλλά το παρουσιάσατε ως απόρρια ενός καλού διατροφικού προγράμματος είναι αληθές αυτό, αλλά είναι και η αιτία του. Αν θέλουμε να δούμε τις υφέρπουσες αιτίες, θα πρέπει να δούμε ότι στη δημογραφική αυτή ανάπτυξη ε, υπήρξαν συνέπειες. Θα δεχτούμε λοιπόν ότι και αυτό ήταν μία, είναι μία αιτία της φτώχειας, κάτι το οποίο δεν έχουμε κάνει μέχρι τώρα. γιατί πολλοί πιστεύουν ότι ε, δεν πρέπει να παρέμβουμε. Από τότε που είπε ο Πάπας δύο παιδιά να οικογένεια, πιστεύω, θα πρέπει να μας απασχολήσει και μας αυτό. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν πρέπει να το θίξουμε για θρησκευτικούς λόγους. Επίσης, η αντιπρόεδρος μας μίλησε για την αναδάσωση. Οι καλύτεροι δασοκόμοι μας λένε ότι μπορούμε να φυτέψουμε παντού αρκεί να είναι το κατάλληλο έδαφος. Δεν υπάρχουν φιλόδοξα προγράμματα όμως από ό,τι βλέπω στο ύψος των ε, περιστάσεων με βάση τις ανάγκες της ε, δασοκομείας για να κάνουμε κάτι. Δεν υπάρχει ολιστική στρατηγική. Τι αναμένεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα στα πλαίσια ενός νέου τρόπου χρηματοδότησης για την επόμενη επταετία. 2021-2027 δηλαδή. Ο κύριος Πέτερλε είναι εδώ. Έχουμε ασχοληθεί με θέματα υγείας στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και χαίρομαι που βρίσκεστε εδώ. Ευχαριστώ Λίντα και ευχαριστώ κύριε Μπίσλε γιατί μας μιλήσατε για τις σκέψεις σας και την πείρα σας. Βεβαίως η Σαχάρα όλο ένα και διευρύνεται, κάτι το οποίο έχει σημαντικές συνέπειες όπως γνωρίζουμε όλοι. Θα ήθελα να σας συγχαρώ για αυτή την απλή ε, μέθοδο που είναι αποτελεσματική των ημισελήνων. Δεν χρειαζόμαστε νέα χρήματα για έρευνες, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη γνώση που προϋπάρχει. Θα ήθελα Ε, εμείς ως εταίροι να καλύψουμε και τις δύο πτυχές, να είναι ένας επίτροπος δηλαδή που θα ε, ασχοληθεί με τα ανθρωπιστικά ζητήματα και τα αναπτυξιακά. Γιατί πολλές φορές δεν χρειαζόμαστε περισσότερα χρήματα, αλλά μία καλύτερη ενιολογική στήριξη των προγραμμάτων η κυρία Ζόφκο. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Διευθυντά, σας ευχαριστούμε που βρίσκεστε εδώ. Ήξερα τον προκάτοχό σας σε περίοδο κρίσης στη Σύρια. Τότε ήμουνα στη Ρώμη. Μπορείτε να μας εξηγήσετε κάπως αυτές τις δυσκολίες που υπάρχουν της προσέγγισης των ΙΠΑ ε, ως προς την πολυμερή προσέγγιση. Πώς το αντιμετωπίσετε, γιατί εσείς ε, ήρθατε σε επαφή και με τους πρέσβεις στη Ρώμη. Ως προς την κρίση στην Ιεμένη, πώς βλέπετε την κατάσταση να εξελίσσεται μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Ιεμένης. Πώς θα επηρεάσει την κατάσταση στην Ιεμένη. Σας επενώ για όσα έχετε κάνει. Είναι εξαιρετική η εργασία σας, ιδιαίτερα επενετέα και σας ευχαριστούμε πολύ. Άλλες ερωτήσεις, όχι. Ε, νομίζω ότι καλύψαμε ένα ευρύ φάσμα. Ωραία, θα προσπαθήσω να συνοψίσω. Καταρχήν σε σχέση με ε, την τεχνολογία εμείς της είπα, είμαστε ο μεγαλύτερος ε, χρήστης των ε, drones, των δορυφορικών συστημάτων, των blockchains και πιστεύουμε ότι αυτό το λογισμικό μπορεί να μας εξοικονομήσει 100 εκατομμύρια δολάρια ετησίως με βάση τα blockchains που αναπτύσσουμε στις βάσεις δεδομένων. Κάτι που με ικανοποιεί είναι το εξής. Εάν μπορούμε να εξοικονομήσουμε 25 σέντ, τότε έχουμε ένα γεύμα για τα παιδιά. Στο Νότιο Σούδαν, μέσα στα πλαίσια των νέων εξελίξεων, στέλαμε με ελικόπτερα φαγητό Δηλαδή ε, είχαμε αυτές τις ρήψεις φαγητών με τα ελικόπτερα. Ε, και φυσικά τα ε, έλαια μαγειρέματος δεν μπορούσαμε να τα ρίξουμε από τον αέρα. Γι' αυτό εμείς αναπτύξαμε ένα νέο σύστημα αλεξίπτωτου όπου δεν χρειαζόταν να βάλουμε το φαγητό ή το λάδι στα ελικόπτερα και μετά να γίνει η ρήψη αυτή η νέα τεχνολογία των ε, αλεξίπτωτων και των συμπιεσμένων αυτών ε, πακέτων στο Νότιο Σουδάν μας οδήγησε σε εξοικονόμηση 25 εκατομμυρίων δολαρίων. Θέλουμε την καινοτομία. Στην, ε, στο Μόναχο με τον επιταχυντή, με το πρόγραμμα του επιταχυντή που χρηματοδοτούμε, προσπαθούμε να δούμε ποιες ιδέες μπορούμε να προωθήσουμε. Αν δεν είναι υψηλής ε, κλίμακας, τότε το κλείνουμε. Ε, αυτό αφορά και την βιοπικιλότητα. Γίνονται πολλές ε, μελέτες μέσα στα πλαίσια του hydroponics και προσπαθούμε και στην Αλγερία και αλλού να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Αυτό αφορά όλους τους προσφυγικούς καταβλισμούς. Ως προς το σύστημα Alibaba, στο Songho είχαμε μία συνάντηση δυόμιση εβδομάδες ε, πριν, αφού άφησα τους ε, Ροχίνια, παρευρέθηκα στην Κίνα, γιατί θεώρησα ότι θα πρέπει και ο ιδιωτικός τομέας να συμμετάσχει και στα πλαίσια της τεχνογνωσίας. Και είπα στον ιδιωτικό τομέα, δεν με, ε, δεν με ενδιαφέρει το χρήμα σας, αλλά η στρατηγική σας συμμετοχή για να αντιμετωπίσετε τη φτώχεια. Έτσι λοιπόν ε, συμμετείχαμε σε πληθώρα μέσων. Επίσης συζητούμε με μεγάλες ε, αγροτικές επιχειρήσεις για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα στις χώρες. Δεν θέλω τα χρήματά σας, τους λέω, θέλω την πραγματογνωμοσύνη σας. Αυτές οι μεγάλες επιχειρήσεις θέλουν να μπουν και να έχουν ένα υψηλό κέρδος από την επένδυσή τους. Βεβαίως, ας έχουν κέρδος, αλλά φέρουν και κοινωνική ευθύνη. Και θεωρώ ότι οι επενδυτές σας θα σας υποστηρίξουν. Αν πείτε σε μια χώρα έχετε λίγο χαμηλότερο κέρδος, αλλά σταθεροποιήστε μια φτωχή χώρα στον κόσμο. Και έτσι οι εκπατριστέντες να μπορέσουν να ενσωματωθούν δηλαδή να υπάρχει μία βιωσιμότητα. Είχαμε λοιπόν πολλές συζητήσεις επί του θέματος ως προς τους σπόρους, καλύτερη σπόρη, καλύτερη τεχνολογία, καλύτερη επένδυση. Αυτό είναι ένας κρίσιμος τομέας, γιατί περνάμε από τον ανθρωπιστικό τομέα όπου δίνουμε αγαθά ή κάνουμε ταμιακές μεταφορές Πολλές φορές δεν μπορεί να γίνει μια τέτοια ταμιακή μεταφορά. Πρέπει να δοθούν αγαθά. Γι' αυτό αξιολογούμε την κάθε κατάσταση. Η κατάρτιση όμως είναι πολύ σημαντική. Χορηγούνται χιλιάδες εκατομμύρια δολάρια έτσι ώστε να επεξεργαστούμε νέα συστήματα διατροφικής αλυσίδας. Ζητώ λοιπόν από τους δωρητές και οργανισμούς να χρησιμοποιήσουν εμάς γιατί μπορούμε να δώσουμε πολλαπλάσιο κέρδος και δεν μας ενδιαφέρει ε, να επενέσουν εμάς, θέλουμε να προωθήσουμε τη βιωσιμότητα. Ως προς τη διατροφική ασφάλεια είναι κρίσιμο το ζήτημα. Εάν δεν το αντιμετωπίσουμε έμπρακτα, δεν θα καταφέρουμε τίποτα. Γι' αυτό τα Ηνωμένα Έθνη πέρασε αυτό το ψήφισμα που λέει ότι η διατροφική ασφάλεια είναι κρίσιμη για την σταθερότητα και την ειρήνη ανά το κόσμο. Αναγνωρίζεται λοιπόν αυτό και θα κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Σε ορισμένα σημεία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τεχνολογία, την τεχνολογία, υψηλή τεχνολογία και να προωθήσουμε τον προγραμματισμό με βάση και τις κλιματικές αλλαγές. Αλλά σε ορισμένα σημεία χρειάζονται λύσεις του 16ου αιώνα. Χρειάζονται δηλαδή πρακτικές λύσεις που να λειτουργούν σε κάθε χώρα χωριστά. Ό,τι, ό,τι λειτουργεί στον Νίγηρα δεν λειτουργεί στην Ιεμένη. Γι' αυτό θα πρέπει να βρούμε τον καλύτερο τρόπο για την κάθε χώρα. Δεν ξέρω ποιος είπε, αλλά ε, η Γερμανία έχει ένα πρόγραμμα εδώ, το Ηνωμένο Βασίλειο εκεί ή παλού, αλλά δεν υπάρχει αλληλοβοήθεια. Κάποιος μου είπε ότι «David, θα πρέπει να υπάρχει επιτόπια συνεργασία από όλους». Μα ναι, εγώ χρειάζομαι από εσάς τη συνεργασία, γιατί οι χώρες της δύση θα πρέπει να προωθήσουν την συνεργασία τους επιτοπίως να υπάρχει μία συνεκτική, ολιστική προσέγγιση από τις ε, δυνάμεις ε, της δύση. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Ένα πρόγραμμα στο Αφγανιστάν. Ιστορικά, στο Μαζάρ Ελσαρίφ ε, ρίχναμε τρόφιμα. Ωραία. Έτσι λοιπόν δεν γινόταν στράτευση των Ταλιμπάν. Αλλά εμείς δεν θέλουμε μόνο τη ρήψη τροφίμων. Μπορούμε να στείλουμε χρήματα, να έρθουμε σε επαφή με τους αγρότες που να χρησιμοποιήσουν τους πόρους ε, για συγκεκριμένες καλλιέργειες και έτσι εμείς αγοράζουμε τους πόρους σε μια συγκεκριμένη τιμή, αυτή είναι η ποιότητα που θέλουμε και έτσι γίνεται η αγορά. Άρα οι αγρότες ε, έκαναν περισσότερες, περισσότερες προσλήψεις, αγόρασαν περισσότερα ε, φορτηγά, προωθήσαμε την τοπική οικονομία αγοράζοντας τους πόρους από το συγκεκριμένο μήλο. Και μετά έγινε η μεταφορά στην περιοχή Μαζάρελ Σαρίφ και τους είπαμε θα σας δώσουμε τρόφιμα υπό τον όρο ότι θα μας βοηθήσετε να διαμορφώσουμε το αγροτικό τοπίο, δηλαδή μιλάμε για μία περιοχή 50.000 εκταρίων. Εάν, υπήρχε, εάν δεν υπήρχε βροχή θα ερχόταν ξηρασία, γιατί πρόκειται για ημιορεινή περιοχή. Δηλαδή, τους βοηθήσαμε να αναδιαμορφώσουν την ορεινή αυτή περιοχή με αρδευτικά έργα, με πηγάδια, με υδροδότηση, με τεχνητές ε, λίμνες και ούτω καθεξής. Και τώρα μου λένε ότι τα παιδιά μας δεν μεταναστεύουν, δεν μπαίνουν στις δυνάμεις των Ταλιμπάν, ζουν στη χώρα τους. Δηλαδή το ίδιο δολάριο το μεγιστοποιήσαμε, μεγιστοποιήσαμε την απόδοσή του ανθρωπιστικά. Αυτά είναι τα προγράμματα που θέλουμε να προωθήσουν και ε, σε περιπτώσεις που δεν πηγαίναν τα παιδιά στο σχολείο, εγώ είπα ας προωθήσουμε τα σχολικά ε, συσίτια. Στο τσάντ όλα αυτά. Δηλαδή, ε, με βοήθησαν οι γυναίκες και στη συνέχεια τα παιδιά πηγαίναν στο σχολείο. Δηλαδή οι μητέρες προώθησαν αυτή την αλυσίδα, οι οποίες καλλιέργησαν 10 εκτάρια για προϊόντα για τα παιδιά. Το 1 τρίτον πάει προς τα παιδιά που πηγαίνουν στο σχολείο εκείνη την ημέρα. Το 1 τρίτον επιστρέφει με τα παιδιά στο σπίτι για να καταναλωθεί ε, εκεί και το άλλο τρίτο το προωθούν οι μητέρες στις αγορές να πουληθεί και να δοθεί στους δασκάλους. Δηλαδή, μου είπαν ότι αν έχουμε 20 εκτάρια και όχι 10 θα είμαστε απόλυτα βιώσιμοι στη ε, Σομαλία, στην Αιθιοπία. Επίσης προωθείται ένα παρόμοιο πρόγραμμα με 75.000 δολάρια. Ως προς τη χρηματοδότηση των ΗΠΑ και τις πολυμερείς σχέσεις στην Ουάσιγκτον προώθησα πολύ, ε, πολλές συζητήσεις, δαπάνησα πολύ χρόνο με το UNHCR, τη UNICEF, αυτούς τους οργανισμούς με τους οποίους εργαζόμαστε καθημερινά. Υπάρχει λοιπόν πολυμερής βοήθεια. Μην βλέπουμε μόνο τα αρνητικά, υπάρχουν και πολλά θετικά και πιστεύω ότι και ο Λευκός Οίκος ε, και το State Department και οι Ρεπουμπλικανοί και οι Δημοκράτες θέλουν να προωθήσουν αυτό το ζήτημα. Ας μην αφήσουμε το δέντρο να μας κρύψει το δάσος. Και θα παραμείνω εδώ. Πριν σας ε, αποχαιρετήσουμε. Θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας πει ποιες είναι οι ιδέες που θέλει να προωθήσει. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα <clears throat> επιθυμώ να πω πόσο πολύ ε, αξία αποδίδουμε στη συνεργασία μας με το WFP που είναι ο νούμερο ένα εταίρος μας σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση που οδεύει από το ΕΚΟ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το WFP και αν εξετάσετε και πόσο πολύ και συνεργαζόμαστε πάρα πολύ στενά, παρόλο που έχουμε δύο επιτρόπους ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συνεργαζόμαστε πάρα πολύ στενά με του συναδέλφου μα, τη ΔΕΒΚΟ, της ε, Αναπτυξιακής συνεργασία. 1,2 δισεκατομμύρια δώσαμε το 2017 μαζί και οι δυο. Αν συμπεριλάβετε και τις ε, ε, συνεισφορές των χωρών μελών, φτάνουμε τα 3 δισεκατομμύρια. Δηλαδή στην ουσία βάλαμε και λεφτά και καλύψαμε λεφτά και αυτά που λέμε. Δεν είναι μόνο υποσχέσει δηλαδή. Σε ό,τι αφορά την Ιεμένη, εδώ πραγματικά δεν θέλω να πω σε περισσότερε λεπτομέρειε γιατί πολλά ήδη εξηγήθηκαν. Λίγα πράγματα μόνο. Πρώτα, είναι στην ημερήσια διάταξη σήμερα της του... του Συμβουλίου Εξωτερικών η ανθρωπιστική κατάσταση στην Ιεμένη που ασφαλώς υπογραμμίζω και εγώ ότι επιδεινώνεται συνεχώς και θέλω να συγχαρώ με την έννοια αυτή και να συγχαρώ τον WFPO διότι είναι πάρα πολύ σημαντική η ανταπόκριση του. Όχι μόνο υλοποιούμε τις δεσμεύσεις αλλά και επικοινωνούμε με ταξί μας και με αυτούς επιτόπου και ο ένας οργανισμός με τον άλλο. Ο δε Επίτροπος Τηλιανίδης προ λίγων ημερών ανακοίνωσε πρόσθετα 90 εκατομμύρια ευρώ υπέρ της Ιεμένης ως ανταπόκρισή μας στις πρόσθετες αυτές ανάγκες και συνεργαζόμαστε πάλι με το WFP για διάφορους ε, τρόπους χορήγησης και μετρητών με διάφορα βάουτσερ, με ε, πίστοση χρεωστικών καρτών κλπ. Και συμφωνώ με τα όσα είπατε σχετικά με το πώς να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της ρευστότητας από τη μια μεριά, αλλά από την άλλη μεριά να χρησιμοποιηθεί παν διαθέσιμο μέσον για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση επιτόπου. Μία πρόσθετη προφορία σχετικά με την Εμένη που νομίζω ότι είναι σημαντικό να τονιστεί είναι ότι πάνω από το μισό διεθνές ανθρωπιστικό προσωπικό που υποτίθεται ότι θα έπρεπε να είναι στη χώρα είναι εκτός και περιμένει τις προξενικές θεωρήσεις. Όταν μιλούμε για ανταπόκριση λοιπόν πρέπει με κάποιον τρόπο να λέμε και όλα τα γεγονότα, το τι συμβαίνει δηλαδή. Θα μπορούσαμε ενδεχομένω να κάνουμε πολύ περισσότερα και πάντως πολύ καλύτερα στην Ιεμένη εάν η το ανθρωπιστικό προσωπικό δηλαδή μπορούσε να είναι επιτόπου και το προσωπικό των δωρητών. Η γεμενήτικη κυβέρνηση δεν δίνει προξενικές θεωρήσεις ήδη από τον Ιούλιο του 2018 και είμαστε στο Νοέμβριο. Αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντική υπόθεση. Θα ήθελα επίσης να πω λίγα λόγια για την Σαχέλ. Ο κύριος Μπίσλεϊ τα είπε βέβαια. Θέλω να πω για το Τσάντ. Πρόσφατα πέρασαμε από εκεί με αποστολή μαζί με τον εκτελεστικό διευθυντή σας ή διευθυντή σας Ντενής, με τον ΦΑΟ, με τη UNICEF και με την Παγκόσμια Τράπεζα. Για να πάμε επί τόπου όλοι μαζί και να δούμε τι ακριβώς πρέπει να γίνει. Και στην χώρα αυτή, Τσάντ, ο αριθμός παιδιών με σοβαρό υποσυτισμό φτάνει σε 300.000 και 2 εκατομμύρια άνθρωποι χρειάζονται επισυτιστική βοήθεια. Και δεν μιλούμε μόνο για σύγκρουση, βεβαίως η σύγκρουση επηρεάζει το Τσάντ, αλλά είναι και τα αποτελεσμάτα της κρίσης στη Λιβύη Υπάρχουν οι πρόσφυγες στο Τσάντ, υπάρχει οικονομική κρίση. Με απεργία των δημοσίων υπαλλήλων. Αν φύγει από την Τζαμένα που είναι η πρωτεύουσα δεν βλέπει τίποτα. Δεν υπάρχει απολύτω καμία παρουσία του κράτους στην υπόλοιπη χώρα. καταστάσεις όπως το Τσάντ αλλά και όλη στην Σαχέλ που είπε κιόλα ότι βρίσκεται σε μια πραγματική κρίση και πολύ σωστά. Είναι κάτι τι που θέλουμε να αντιμετωπίσουμε μαζί σας. Ναι, ναι, θα, θα, θα ολοκληρώσω αμέσως. Γίνονται πολλές συζητήσεις για τη σχέση ανθρωπιστικής βοήθειας με αναπτυξιακή. Σε πολλές από τις χώρες ΑΧΕΛ ξεφεύγουμε πια από την αναπτυξιακή βοήθεια και επανερχόμαστε στην ανθρωπιστική. Η κλιματική αλλαγή είναι και αυτό μια θεμελιώδης πτυχή της καταστροφής. Αν μου επιτρέψει μια φράση για τον Μπαγκλαντές. Κάνουμε πάρα πολλά μαζί. Πρέπει να δώσουμε και περισσότερα στο τμήμα της ρευστότητα, δηλαδή της χορήγησης ρευστού και ναι, λίγο λιγότερο από δύο χρόνια. Ε, είναι προφανές ότι έχει φέρει πολύ πάθος και αφοσίωση στο World Food Program. Θα επανέλθουμε, θα πάμε και στην Τουρκία του χρόνου. Ευχαριστώ πολύ. Τηρείτε τις δεσμεύσεις των Εθνών για το πρόγραμμα. Θα προσπαθήσουμε και εμείς από τη δική μας πλευρά να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Σας ευχαριστώ που ήρθατε σήμερα εδώ και να ξανάρθετε. δεν Sorry, can, can people who are leaving at uh, the back... Να ζητήσω από τους συναδέλφους και τους συνεργάτες τους που φεύγουν από το, την αίθουσα να το πράξουν αυτό ήσυχα και όσο το δυνατόν γρηγορότερα για να συνεχίσουμε. Συνεχίσουμε με το σημείο 8 της σημερινής διάταξης, την ενίσχυση τη εταιρική σχέση Ευρωπαϊκή Ένωση Αφρική. Έχουμε αυτό στην ημερησία μεταξύ μα σήμερα. Γνωρίζουμε από την ομιλία για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Πρόεδρου Juncker, ο οποίος ανακοίνωσε για την νέα σχέση τη ευρωπαϊκή ένωση με την Αφρική και την σημασία που έχουν αυτέ οι στρατηγικές. Το επανέλαβε αυτό ο Πρόεδρος Ταγιάννη στην Ολομέλεια, τη σημασία που αποδίδουμε στην σχέση με την Αφρική και η καγκελάριο Μέρκελ όταν μίλησε στην Ολομέλεια αναφέρθηκε στη σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αφρικής. Θα μιλήσουμε σήμερα, θα έχουμε αυτή τη συζήτηση τη βάση αυτών των δύο ανακοινώσεων της Επιτροπής. Θα κάνουμε έναν απολογισμό, θα δούμε πώς εξελίσσονται τα νέα προγράμματα τα οποία προετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την Αφρική. Ε, θα έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Κουντούν και την κυρία Μαρία Ταγέγκερ. Έχουμε και παλαιότερα, είχαμε και παλαιότερα την ευκαιρία να μιλήσουμε με αυτού. Αναπληρωτέ διευθυντέ στην Γενική Διεύθυνση ε, Αναπτυξιακή Συνεργασία και έχουμε επίση και εκπρόσωπο ε, τη Υπηρεσία Εξωτερική Δράση. Ο Κουντούνς, ο κύριος Κουντούνς που θα μιλήσει πρώτος, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, θα είμαι σύντομος γιατί δεν έχετε και πολύ χρόνο στη διάθεσή σας. Πρώτα όλα για τις ανακοινώσεις της Επιτροπής. Όπως αναφέρατε, συνεχίσουμε να θεωρούμε σημαντική ήπειρο την Αφρική. Αυτό, ε, ε, η σημασία της ήπειρο αυτής να γνωρίζεται όλο και περισσότερο. Οργανώθηκε σύνοδος κορυφής στην οποία υιοθετήθηκε η δήλωση της ε, διακήρυξη της Αμπιτζάν του και την οποία θα πρέπει να εφαρμόσουμε στην πράξη. Όλα αυτά έχοντας βεβαίως ε, υπόψη μας τους αναπτυξιακούς στόχους και την προσπάθεια και των δύο πλευρών να, δώσουμε, να εξυγχρονίσουμε την ε, σχέση μας. τη στιγμή γίνεται μια προσπάθεια να μεταφραστεί σε πρακτικούς όρους το μνημόνιο κατανόησης ε, για την ε, ειρήνη και τη διακυβέρνηση και μετά να δούμε το σκέλος της διακήρυξης του Αμπιτζάν για την αναπτυξιακή συνεργασία. Θεωρούμε ότι πράγματι έχει έρθει ο, χρόνος να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση σε αυτό το ζήτημα της ανάπτυξης και ιδίω ένας κύριος στόχος ε, που είναι η δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την Αφρική ως Ήπειρο, για τον πληθυσμό της Αφρικής. Η δημιουργία θέσεων απασχόλησης είναι το σημείο έναρξης και μέσο για την επίτευξη αυτού του στόχου θα είναι οι επενδύσεις. Και αυτό γιατί διαπιστώνουμε σε διάφορες μελέτες που έχουν δημοσιοποιηθεί τους τελευταίους μήνες ότι υπάρχουν τεράστιες ευκαιρίες στην Αφρική, ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον, ότι υπάρχει δυναμική και υπάρχουν επίσης και ευκαιρίες χρηματοδότησης. Μέσω των επενδύσεων η Αφρική θα μπορέσει να δημιουργήσει περισσότερη προστιθέμενη αξία ε, και να βελτιώσει την οικονομία της με τρόπο που θα, θα ωφελήσει τους πολίτες της Αφρικής, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τους. Δεν μιλούμε εδώ για πολυεθνικές από το εξωτερικό. Θέσεις εργασίας λοιπόν και επενδύσεις και μετά έχουμε παρέμβαση σε δύο παιδεία, πρώτα απ' όλα βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και το οποίο μας οδηγεί αμέσω αμέσως στα ζητήματα του κράτου δικαίου, της αντιμετώπισης της διαφθοράς, της διακυβέρνησης, της βελτίωσης της λειτουργίας των θεσμών των κρατών και δεύτερο τομέα, πολύ σημαντικό, που είναι η αντιμετώπιση των κινδύνων γιατί παρά τις διάφορες πρωτοβουλίες θα συνεχίσουν να υφίστανται κίνδυνοι. Το ερώτημα λοιπόν είναι πώς μπορούμε να παρέμβουμε για να τους αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά, ιδίω στις περιπτώσεις εκείνες που εξαιτία των κινδύνων δεν γίνονται επενδύσεις και δεν δημιουργούνται θέσεις απασχόλησης. Κάτι ακόμα το οποίο θα μας απασχολήσει είναι το ζήτημα το, της εξέλιξης των τοπικών οικονομιών, δηλαδή των υπηρεσιών θα χρειαστεί μεγαλύτερη ενσωμάτωση, ενοποίηση μάλλον των τοπικών ε, οικονομιών και επίσης σε επίπεδο υπήρου της αφρικανικής οικονομίας. Και τέλος, είναι πολύ σημαντικό για να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης να είναι έτοιμο και το ανθρώπινο δυναμικό. Και έτσι ερχόμαστε στο, στην τρίτη μας παρέμβαση που θα, θα εστιαστεί στην κατάρτιση, στην εκπαίδευση, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στόχος όλων αυτών των προσπαθειών είναι να έχουμε ουσιαστικά αποτελέσματα επιτόπου συνδυάζοντας αυτές τις προσπάθειες. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Πριν από 10 ημέρες βρισκόμουν στο Ιωάννεσπουργκ επί μια εβδομάδα και παρακολούθησα την, το φόρουμ επενδύσεων στην Αφρική που οργάνωσε η Αφρικανική ε, τράπεζα Επενδύσεων και ένα πάνελ αφορούσε το Τογκό. Μια χώρα όπου ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα είναι ο εξηλεκτρισμός της υπαίθρου. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να δημιουργηθούν σχολεία, μπορεί να δημιουργηθούν νοσοκομεία, μπορεί να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον στο οποίο να αναπτυχθούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις με τον εξηλεκτρισμό. Υπάρχει ενδιαφέρον από τον ιδιωτικό τομέα. Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί δηλαδή η άμεση αναπτυξιακή ενίσχυση για να χρηματοδοτηθούν τέτοια προγράμματα. Υπάρχουν ήδη ε, επιχειρήσεις επιτόπου που ενδιαφέρονται. Η Αφρικανική Αναπτυξιακή Τράπεζα είναι διατεθειμένη να δώσει δάνεια. Παραμένει όμως ένας κίνδυνος. Και εδώ παρεμβαίνουμε εμείς, θα μιλήσει περισσότερο η συνάδελφος. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα σύστημα με το οποίο να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε είτε έναν υφιστάμενο είτε ε, κίνδυνο είτε έναν κίνδυνο ο οποίος απλώς θεωρείται ότι υπάρχει. Αυτό θα έλεγα ότι είναι η περιπτουσία της ε, ανακοίνωσης της Επιτροπής για την ε, για την Αφρική. Ε, τα περισσότερα ήδη ελέγχθησαν. Μιλάμε για εργασία και επενδύσεις. Εγώ ε, επέστρεψα από την αποστολή μου. Θα θυμόσαστε, μιλήσαμε για την διαδικασία του άρθρου 11, Λίντα. Δηλαδή, εγκρίναμε την θέση μας και σήμερα μπορώ να σας πω ότι φτάσαμε σε καλή γνωμοδότηση για τα 30 pips και το 1,5 δις εγγυήσεων. Και υπάρχει θετική γνωμοδότηση. Τώρα είμαστε στη συμβατική φάση έτσι να, έχουμε, να φτάσουμε στις ε, συμβατικές συμφωνίες. Δηλαδή μας ενδιαφέρει να χρησιμοποιήσουμε την επιτυχία του EFSD και να δούμε πώς μπορούμε να προσελκύσουμε τον ιδιωτικό τομέα μαζί με την Αφρικανική Συμμαχία έτσι ώστε να έχουμε καλύτερες επενδύσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα καλύτερο οικοδόμημα και μπορώ να σας πω ότι θέλουμε από δις να φτάσουμε σε τρεις. Αυτός να είναι ο αριθμός με τη συμμετοχή και του ιδιωτικού τομέα. Θα πρέπει επίσης να υπάρχει ο μέγιστος αντίκτυπος χωρίς να περιοριστούν οι πόροι. Άρα η επένδυση παίζει πολύ σημαντικό ρόλο για τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Και εδώ ε, δεν εννοώ μόνο δανειοδότηση αλλά και προσθετικότητα με βάση δηλαδή τη, χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό μας, με βάση την πείρα μας και την, ε, τα συμφέροντα των IFI, φτάσαμε σε 3,5 ε, δις για εγγύηση 1,5 και έτσι θα μπορέσουμε να επεκτείνουμε την εγγύηση και τις επενδύσεις για να δούμε πώς με βάση το παρόν οικοδόμημα μπορούμε να έχουμε καλύτερη χρήση και να είμαστε ε, σε θέση να μιλήσουμε για τις επιπτώσεις. Είχαμε το πρώτο σεμινάριο τον Ιανουάριο, το δεύτερο τον Οκτώβριο και θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την ενεργό συμμετοχή του αυτό είναι δηλαδή και ο στόχος να μεγιστοποιήσουμε τις επενδύσεις στις τρίτες χώρες και να έχουμε και την εξωτερική πλατφόρμα επενδύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι είδαμε κατά τη διαδικασία του EFSD ότι το ανοιχτό αυτό οικοδόμημα επαυξάνει την ποιότητα και γι' αυτό θα θέλαμε να προτείνουμε μία βραχυχρόνια προσαρμογή για τις εξωτερικές επενδύσεις που θα υποστηρίξει ο Ευρωπαϊκός Προϋπολογισμός με βάση τους στόχους που έχουν οριστεί από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, επίπτωση λοιπόν, επιπτώσεις και φυσικά συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Δεν θα ήθελα να σας μιλήσω για ολόκληρη την ανακοίνωση, μπορείτε να τη διαβάσετε. Έχει σημασία τα τρία επίπεδα. Καταρχήν, οι κατευθυντήριες γραμμές για το πολιετές πρόγραμμα χρηματοδότησης. Δεύτερον, η Επίτροπη εγκρίνει το Ταμείο Εγγυήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης έτσι ώστε να μην κάνουμε επικάλυψη, δηλαδή να υπάρχει εξωτερική ανάθεση, όπως κάναμε και στα, με τα EFSD. Και στη συνέχεια να φτάσουμε στις συμφωνίες εγγύσεων και φυσικά να βασιστούμε στην Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή και τις Εθνικές Τράπεζες για συνεργασία. Όπως σας είπα, έχει μεγάλη σημασία και η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα. Με ευχαρίστηση να απαντήσω στις τυχόν ερωτήσεις σας. Η Μαρία Χόιμπουκ ζήτησε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Αν θέλετε φορέστε τα ακουστικά σας για να καταλάβετε, θα μιλήσω γερμανικά. Yeah, σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ για ε, τα όσα εξηγήσατε και ιδίως είπατε ότι θέλετε αυτούς τους τέσσερις πυλώνες της συμμαχίας με την Αφρική να τους συνδέσετε μεταξύ τους. Εμένα με ενδιαφέρει όμως μια άλλη διασύνδεση. Εδώ έχουμε αυτή τη νέα συμμαχία με την Αφρική. Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Γιούνκερ την ανακοίνωσε. Αυτή λοιπόν έχει ξεκινήσει ήδη και προχωρεί εξ όσων ακούω. Αυτό που με εκπλήσει ωστόσο είναι το εξής, διότι Μόλις αρχίσαμε με τις διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία μετά την Κοτονού. Αυτές οι δύο διαδικασίες πώς συνδέονται μεταξύ τους. Μιλήσατε, ότι θέλετε να προωθήσετε την περιφερειοποίηση των σχέσεων ΑΚΕ, αλλά έχει ήδη εγκριθεί ένα συνολικότερο πλαίσιο. Με εκπλήσει το ότι προωθείτε ένα νέο πρόγραμμα, ενώ όπως είπα Μόλις άρχισαν οι διαπραγματεύσεις για μετά την Συμφωνία Κοτονού, μετά την περίοδο μετά την Κοτονού. Άρα προστίθεται μια τρίτη διαδικασία, δηλαδή εμείς συνεχίζουμε να διαπραγματευόμαστε για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Τι θα γίνει στο μέλλον με τα χρήματα και με τα νέα εξωτερικά μας εργαλεία πολιτικής όπως το NDICI και υπάρχουν και εθνικές προσπάθειες όπως αυτό το εντό εισαγωγικών σχέδιο Marshall για την Αφρική από πλευρά Γερμανία. Βλέπω λοιπόν να κινούνται εκ παραλίλου διάφορε διαδικασίε. Στι διαπραγματεύσει όμω, τι γίνεται. Άκουσα κιόλα, ίσω να το έχετε ακούσει κι εσεί, ότι η Αφρικανική Ένωση αποφάσισε να βγάλουν αυτό το α από το ACP, από την Αφρική Καραϊβική Ειρηνικό. Επομένως φαίνεται πως από την Αφρική υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για μια πιο άμεση σχέση με την Ευρώπη. Όλα αυτά τι επιπτώσεις έχουν στις διαπραγματεύσεις. Ο δε Επίτροπος κ. Μίμητσα πώς θα τα μεταφέρει αυτά στις διαπραγματεύσεις. Πρόεδρος Μακ Άβαν. Έχουμε ερώτηση από την αντιπρόεδρό μας, την κυρία Καπέιβα. Ευχαριστώ αγαπητή Πρόεδρε. Μεγάλη ικανοποίηση αισθάνθηκα που άκουσα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Αφρική ε, προχωρούν σε νέα συμμαχία και σε νέα σχέση μεταξύ των και επενδύουν και δημιουργούν απασχόληση. Το βρίσκω θαυμάσιο αυτό. Πολύ καλά κάνουν. Αλλά έχω μια ερώτηση. για τις παλαιότερες και σημαντικές εξελίξεις στον ανθρωπιστικό τομέα, στον ε, τομέα. Τι γίνεται, στον ανθρωπιστικό μάλλον τομέα. Κάνουμε νέα βήματα στην Αφρική και ξεχνούμε τα παλαιά. Ελπίζω όχι. Πώς διαμορφώνεται η κατάσταση μεταξύ των νέων, μάλλον της νέας πολιτικής ανάπτυξης και της παλαιάς. Έχουμε όμως και το κύριο Γιόνσεν από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικών Δράσεων. Θέλετε να τοποθετηθείτε σύντομα. Τα πιο πολλά λέχθηκαν. Αλλά μετά το Αμπιτζάν συμφωνήσαμε τον Μάιο σχετικά με ένα μνημόνιο συμφωνίας για Peace, Security και Governance που είναι ο πρόδρομος της ε, συμμαχίας που διαμορφώνεται. Αυτό το μνημόνιο συμφωνίας στοχεύει ιδιαίτερα σε θέματα δημοκρατίας, διακυβέρνησης, παρακολούθηση εκλογών, βεβαίως στον τομέα της πρόληψης, γυναίκες, ειρήνη, ασφάλεια κλπ. Και εξετάζουμε πώς μπορούμε να ενισχύσουμε την εφαρμογή του Μνημονίου Συμφωνίας. Αυτά όλα θα ακολουθήσουν την δήλωση Αμπιτζάν και τα τέσσερα σκέλη που συμφωνήθηκαν εκεί από αρχηγού κρατών και κυβερνήσεων και μέχρι την επόμενη διάσκεψη κορυφής και εκεί θα καταγράψουμε την πρόοδο στο υπουργικό επίπεδο που έχει άλλωστε ζητήσει η διάσκεψη κορυφής και που νομίζουμε ότι θα μπορέσει να γίνει αρχή του επόμενου έτους μεταξύ Αφρικανικής Ένωσης και Ευρωπαϊκής Ένωσης για να εξεταστεί η πρόοδος που θα έχει σημειωθεί σε αυτούς τους διαφορετικούς τομείς. Κουν θέλετε εσείς πρώτος να απαντήσετε. Σα ευχαριστώ πολύ. Όσον αφορά πρώτα απ' όλα τι διαφορετικέ διαδικασίε που ακολουθούνται. Μπορεί να δίνει την εντύπωση ότι είναι περίπλοκο το σύστημα, όμω, στην πραγματικότητα δεν είναι. Ξεκινώ με τη Συμμαχία για την Αφρική. Αυτή η συμμαχία προσπαθεί να υλοποιήσει την ατζέντα που, στην οποία συμφωνήσαμε στο Αμπιτζάν μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών της Αφρικής στην κοινή Σύνοδο Κορυφής. Αυτό ήταν το σημείο κίνησής μας και αυτό υλοποιούμε αυτή τη στιγμή με τη μορφή της συμμαχίας. Και όπως είπε και ο το δεύτερο μέρος της διακήρυξης του Αμπιτζάν, αυτό που αφορά περισσότερο στην ασφάλεια και τη διακυβέρνηση, θα ακολουθήσει και θα υλοποιηθεί μέσω του μνημονίου. Από τη στιγμή που θα λειτουργήσει η ε, συμμαχία θα φροντίσουμε η παρέμβασή της να είναι συμβατή και να συνδυάζεται καλά με τις πρωτοβουλίες των κρατών μελών. Αυτό δεν ε, το καλωσόρισαν μόνο οι εταίροι μας από την Αφρική, το καλωσόρισαν επίσης και τα κράτη-μέλη. Δηλαδή φαίνεται ότι τα κράτη-μέλη επιθυμούν να συνεργαστούν μαζί μας για σε αυτό το τομέα. Γιατί βεβαίω είναι προ όφελο όλων να υπάρχει σωστό συντονισμό ανάμεσα σε αυτό που εμεί πράττουμε και αυτό που κάνουν τα κράτη-μέλη. Αυτό θα οδηγήσει σε καλύτερα αποτελέσματα σίγουρα από ότι αν, δεν, αν υπάρχει έλλειψη συντονισμού. Κάτι αντίστοιχο μπορεί να πει κανείς και για το σύμφωνο των G20 για την Αφρική. Ε, ε μια πρωτοβουλία στην οποία είναι ιδιαίτερα δραστήρια ακόμα η Γερμανία. συνδέεται άμεσα με τις δικές μας πρωτοβουλίες για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στις χώρες αυτές. Ναι, υπάρχουν λοιπόν κάποιες παράλληλες πρωτοβουλίες, όμως μέσω της συμμαχίας χτίζουμε και μια πλατφόρμα η οποία θα εξασφαλίζει ότι οι διάφορες πρωτοβουλίες που γίνονται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι συνεκτικές, όχι μόνο αυτές που κάνει η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά επίσης και οι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν και τα κράτη-μέλη προσπαθούμε όλο και περισσότερο να προγραμματίζουμε τις παρεμβάσεις μας από κοινού. Και αυτό με φέρνει στη συζήτηση για το επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Όλες οι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουμε αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο πλαίσιο του τρέχοντος δημοσιονομικού πλαισίου και του τρέχοντος προϋπολογισμού. Βεβαίως έχουμε υποβάλει προτάσεις. και η πρότασή μας ε, σε σχέση με το NDICI θα δείτε ότι υπάρχει πλήρης ε, συνεκτικότητα μεταξύ των πρωτοβουλειών που έχουμε ήδη αναλάβει στο πλαίσιο του τρέχοντος ε, πολιτούς δημοσιονομικού πλαισίου και Τη πρότασή μα για το επόμενο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο που αυτή τη στιγμή συζητούμε με εσά το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Επομένω, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα συνεκτικότητα, Θα έλεγα μάλλον ότι το δεύτερο είναι ε, συνέχεια του πρώτου. Και έρχομαι λοιπόν και στο ερώτημα για τι τις, μετά το Κοτονού και τι διαπραγματεύσει, μάλλον για του στόχου μετά το Κοτονού. Οι διαπραγματεύσει έχουν ξεκινήσει από τα θεμελιώδη στοιχεία να δούμε δηλαδή τι είναι αυτό που συνδέει τις χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού και μετά αφού συμφωνήσουμε σε αυτά τα θεμελιώδη στοιχεία, θα προχωρήσουμε στις διαπραγματεύσεις για τους πυλώνες τους ξεχωριστούς. Ε, βεβαίως, σε σχέση με τον πυλώνα της Αφρικής, το σημείο εκκίνησης θα είναι η διακήρυξη του Αμπιτζάν, γιατί αυτό είναι το σημείο αναφοράς και για την Αφρικανική Ήπειρο και για την ε, ε, ε, Ευρωπαϊκή Ένωση, μιας και είχε διατυπωθεί, είχε διακηρυχθεί αυτή η διακήρυξη από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων. Βλέπετε λοιπόν ότι δεν υπάρχει κάποια σύγκρουση, κάποιο πρόβλημα στο, στο σημείο κίνηση των πρωτοβουλίων που θα αναλάβουμε μετά το κουτουνού ή αυτών που έχουμε ήδη αναλάβει. Το ένα οδηγεί στο άλλο. Με ρωτήσατε επίση για το μέλλον τη ε, λεγόμενη παραδοσιακή αναπτυξιακή βοήθεια. Ε, εγώ πιστεύω ότι αυτέ οι πρωτοβουλίε που αναλαμβάνουμε ουσιαστικά είναι παραδοσιακέ ε, πρωτοβουλίες αναπτυξιακής βοήθειας. Όλες αυτές οι πρωτοβουλίες που θα αναλάβουμε στο πλαίσιο της συμμαχίας ταιριάζουν με αυτές που είχαμε αναλάβει στο παρελθόν και επίσης αποτελούν ουσιαστικό σκέλος μιας πραγματικής ατζέντα για την ανάπτυξη. Αυτό που προσπαθούμε να επιτύχουμε είναι να υπάρχει μεγαλύτερη συνεκτικότητα ανάμεσα στις διάφορες ε, πρωτοβουλίες. Δηλαδή, για παράδειγμα, εάν διαπιστώσουμε ότι σε κάποιον τομέα, σε κάποια περιοχή υπάρχει δυνατότητα να δημιουργηθούν περισσότερες θέσεις απασχόλησης, οι προσπάθειες μας σε αυτό θα πρέπει να ταιριάζουν με τις προσπάθειές μας στον τομέα της εκπαίδευσης. Εάν σωστά ακολουθήσουμε τους στόχους της συμμαχίας, αυτό που θα συμβεί είναι ότι οι προσπάθειες μας για την εκπαίδευση, για την επαγγελματική κατάρτιση και η παρέμβασή μας στην αγορά εργασίας θα οδηγήσουν πραγματικά στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Και αυτό με οδηγεί και στο υπό, επόμενο συμπέρασμα, ότι δεν υπάρχει κάποιο είδους αποχώρηση από παραδοσιακά ζητήματα ενδιαφέροντος, όπως για παράδειγμα την πρόσβαση στο νερό, την βελτίωση των αποχετευτικών συστημάτων. Η υποστήριξή μας προς τις χώρες αυτές θα συνεχίσει να υφίσταται. Το ίδιο ισχύει και για την υποστήριξή μας στα ζητήματα, ζητήματα τα θεσμικά της διακυβέρνησης. Και αυτές οι παρεμβάσεις συνεχίζουν να αποτελούν μέρος της ε, συμμαχίας. Δεν υπάρχει λοιπόν κάποιο είδου ε, υποβάθμιση αυτών των ζητημάτων. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι οι όποιε μα πρωτοβουλίε να είναι καλύτερα συντονισμένε. Βεβαίω θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στην συμπληρωματικότητα των διαφόρων χρηματοδοματικών εργαλείων. Το ίδιο ισχύει και για τη συμπληρωματικότητα που πρέπει να έχουν τα αναπτυξιακά προγράμματα με τα ανθρωπιστικά προγράμματα και την ε, προσπάθεια μας για την πρόθεση της ειρήνης. Θα συνεχιστεί η συνεργασία μας με τους αρμοδίους συναδέλφους στα άλλα τμήματα της Επιτροπής. Η Πρόεδρος Μαρκέβαν, σας ευχαριστούμε. Βεβαίως θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε το θέμα. Γνωρίζω ότι οι συνεισηγητές μας ε, έχουν καταλήξει στο πρώτο προσχέδιο της έκθεσής τους, μεταφράζεται. Θα συνεχιστεί λοιπόν η συζήτηση για το θέμα αυτό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα του εκπροσώπου τη Επιτροπή και τη Υπηρεσία Εξωτερική Δράση για την παρουσία του εδώ και για τι ε, παρουσιάσει που μα έδωσαν για αυτέ τι σημαντικέ πρωτοβουλίε που έχουμε αναλάβει έτσι ώστε να εξυγχρονιστεί η σχέση μα με την Αφρικανική Ήπειρο. Ε, θα πρέπει να σας παρουσιάσω το σημείο 9 και μετά θα δώσω το λόγο στον Ρίκε Γκερέρο, που θα αναλάβει το τελευταίο μέρος της Προεδρίας, γιατί εγώ πρέπει να αποχωρήσω. Λοιπόν, θέμα υπαριθμών 9. Σύσταση προς την ύπατη εκπρόσωπο και το Συμβούλιο σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο για τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό για την Ειρήνη. Είναι στα πλαίσια του, του νέου ΠΔΠ και πρόκειται για μία εκτός προϋπολογισμού χρηματοδότηση από τα κράτη-μέλη για την ειρηνευτική διαδικασία. Ξέρουμε ότι η συνθήκη δεν επιτρέπει καμία χρηματοδότηση η οποία θα μπορούσε να έχει σχέση με την άμυνα. Δηλαδή δεν θα πρόκειται πλέον για APF αλλά για EDF. Άρα το Κοινοβούλιο έχει πολύ περιορισμένες αρμοδιότητες και η ΣΕΝΤΕ, η υποεπιτροπή ΣΕΝΤΕ θα γνωμοδοτήσει. Και για τεχνικούς λόγους, και δεν θυμάμαι καν τους ε, κανόνες, εμείς ως ΔΕΒΕ δεν μπορούμε να γνωμοδοτήσουμε επίσημα προς τη ΣΕΝΤΕ αλλά θεώρησαν οι συντονιστές ότι υπάρχουν σημαντικά στοιχεία που θα πρέπει να τονίσουμε προς την Επιτροπή ΣΕΝΤΕ. Άρα προτείνουμε είτε η πρόεδρος ε, ε, είτε τα μέλη θα μπορούσαν να προωθήσουν τροπολογίες για σημαντικά ζητήματα για τους βιώσιμους στόχους ε, της χιλιετίας και για να τονίσουμε ότι οι αμυντικές δαπάνες δεν θα πρέπει να χρηματοδοτούνται από αυτό τον προϋπολογισμό, αλλά από ένα ξεχωριστό ταμείο. Εμείς το συζητήσαμε στα πλαίσια του ICSP. Αύριο το πρωί θα προτείνω εννέα τροπολογίες που θα ψηφίσουμε ξεχωριστά και νομίζω ότι οι συντονιστές και οι πολιτικές ομάδες είπαν ότι τις υποστηρίζουμε. Μετά θα τις στείλουμε στη ΣΕΝΤΕ και ελπίζουμε να τις συμπεριλάβουν ή τουλάχιστον μερικές από αυτές κατά τη γνωμοδότηση προς το Συμβούλιο. Είναι πολύ σύντομη η έκθεση. Από όσο γνωρίζω, η εκπρόσωπος της ΕΙΕΔ είναι εδώ. Δεν έχω τα ονόματά σας, άρα θα θέλαμε να μας πείτε ποιοι είστε. Ο Ακίν Τάσο είμαι ε, υπεύθυνος ε, για θέματα Αφρικής. Δεν θα μπορέσω να γνωμοδοτήσω για το παρόν έγγραφο, απλώς να σας ε, μιλήσω για τη φύση αυτού του μέσου. Το μέσο αυτό θα συσταθεί με στα πλαίσια της ΕΙΕΔ της ΚΕΠΑ δηλαδή, δεν είναι πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά είναι πρόταση της ΥΠΑ της εκπροσώπου με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι μια δυνατότητα που υπάρχει στη συνθήκη ε, που χρησιμοποιούμε όπως κάτι το οποίο, συγγνώμη, δεν είχε γίνει στο παρελθόν. Πρόκειται για έναν προϋπολογισμό για CFSP τη στιγμή που υπάρχει, υπάρχουν στρατιωτικές επιπτώσεις. Δεν πρόκειται για αναπόσπαστο μέρος του ΠΔΠ, είναι μια παράλληλη διαδικασία, αλλά δεν περιλαμβάνεται στον κοινοτικό προϋπολογισμό. Επίσης, η Ένωση θα πρέπει να έχει τα κατάλληλα μέσα για να αντιμετωπίσει θέματα εξωτερικής πολιτικής, ανάπτυξης, γειτονίας, ανθρωπιστικής βοήθεια ή θεμάτων της ΚΕΠΑ. δεν θα γίνει καμία ε, χρηματοδότηση από το DCI ή καμία αναπτυξιακή πολιτική γιατί θα υπάρχει ένα ξεχωριστό ε, ταμείο από τα κράτη-μέλη. Αυτά είναι τα πλαίσια λειτουργίας, δηλαδή δεν υπάρχει αιτιώδη συνάφεια μεταξύ των δύο. Ευχαριστούμε πολύ. Ωραία. Έχουμε σαφή άποψη ότι όταν μεταβήκαμε στην κεντροαφρικανική δημοκρατία είδαμε ότι πρέπει να έχουμε άλλα μέσα γιατί όλα τα χρήματα που δαπανούμε ε, για ε, στρατιωτικές επιχειρήσεις, η κατάρτιση και ούτω καθεξής δεν ε, μπόρεσε να έχει πλήρη ανταπόκριση και έτσι μπήκαν στη μέση οι Ρώσοι. Άρα Αύριο το πρωί λοιπόν θα ψηφίσουμε και θα στείλουμε τις τροπολογίες της ΣΕΝΤΕ. Λοιπόν, εδώ θα παραμείνουμε και θα δώσω... Θα αναθέσω την Προεδρία στον Ενρίκε Γκερέρο, ο οποίος θα με αντικαταστήσει από το σημείο 10 και υστερότερα. Ευχαριστώ. Εγώ θα σας δω αύριο το πρωί. Τώρα θα προχωρήσουμε σε ανταλλαγή απόψεων στην γνωμοδότησή μας για ένα νέο πρόγραμμα Εράσμους για την εκπαίδευση, κατάρτιση, νεολαία και αθλητισμό. Στόχος αυτού του προγράμματος είναι να αντικαταστήσει το Εράσμους Plus και να δημιουργήσει έναν νέο εκπαιδευτικό χώρο μέχρι το 2025, έτσι ώστε να φτάσουμε πιο κοντά στους ανθρώπους διαφόρων ηλικιών και πολιτισμικού, ε, κοινωνικού και οικονομικού ε, background. Αυτό που έχει λοιπόν σημασία είναι επίσης να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε και τους ε, κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών ανθρώπων με αναπηρίες και μεταναστών. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να εντατικοποιήσουμε την διεθνή κινητικότητα και συνεργασία με τρίτες χώρες, έτσι ώστε να έχουμε ένα νέο μέσο εξωτερικής χρηματοδότησης, NDICI, και θα μπορέσουμε να έχουμε πολυετή ενδεικτικά προγράμματα, αλλά μετά θα εφαρμοστούν μέσω του κανονισμού Εράσμους. Υπάρχουν πολύ περιορισμένες αναφορές ως προς την εξωτερική διάσταση του ε, σχεδίου κανονισμού για το Εράσμους, γι' αυτό και εμείς ε, θα αποφανθούμε. Η επικεφαλής επιτροπή είναι η ΚΑΛΤ, η οποία θα αποφανθεί με ψηφοφορία στις 21-22 Ιανουαρίου 2019. Ο εισηγητή μα για αυτή τη γνωμοδότηση είναι ο Ιγνάσιο Κοράου, στον οποίο και δίνω το λόγο. Έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Πρόκειται για την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ε, κατάρτιση του προγράμματος Εράσμου, για την εκπαίδευση κατάρτιση νεολαία και τον αθλητισμό το νέο πρόγραμμα, έχει μια νέα θεμελιώδη διάσταση η οποία αναφορά, αφορά την κινητικότητα, τη συνεργασία καθώς επίσης και, ε, τέτοιες, ε, και τη διεθνή του διάσταση. Όσον αφορά τη διεθνή του διάσταση, ο στόχος του προγράμματος είναι να υπάρχει συνέργεια μεταξύ των εργαλείων της εξωτερικής δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προώθηση των στόχων της Ένωσης για την προώθηση των θεσμικών μεταρρυθμίσεων και της ανάπτυξης σε τρίτες χώρες. Και στόχο είναι επίση να αξιοποιήσουμε το πρόγραμμα Erasmus για να συνεργαστούμε με την νεολαία αυτών των χωρών, έτσι ώστε να υπάρξει και μεγαλύτερη κατανόηση μεταξύ των διαφορετικών πολιτισμών. Θα έλεγα ότι πρέπει να υποστηρίξουμε αυτή την πρόταση, ωστόσο με ανησυχεί το γεγονό ότι δεν υπάρχουν επαρκεί αναφορέ στη διεθνή διάσταση και πιο συγκεκριμένα στη σύνδεση με των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την εξωτερική δράση με τις ανάγκες των τρίτων χωρών. Πιστεύω ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη οι προτεραιότητε για την αναπτυξιακή συνεργασία όταν θα επιλέγονται οι σχετικοί στόχοι του προγράμματο Εράσμου. Η κυρία Μπιό έχει υποβάλει σχετικές ε, τροπολογίε που συζητήθηκαν και στην προηγούμενη Ολομέλεια. Προτείνω εγώ λοιπόν τροπολογίες με την δική μου έκθεση, έτσι ώστε το προτινόμενο πρόγραμμα να είναι συμβατό με τις αρχές και τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των στόχων εξωτερικής δράσης της, συμπεριλαμβανομένη και της καταπολέμησης της φτώχειας, της συνεισφοράς που θα πρέπει να έχει το πρόγραμμα αυτό στους ε, διεθνείς αναπτυξιακούς στόχους, καθώς επίσης και την συνεισφορά που θα πρέπει να έχει στην εξάλληψη της φτώχειας ε, στις αναπτυσσόμενες χώρες. Αυτό σημαίνει ότι οι διαδικασίες προγραμματισμού θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι το πρόγραμμα θα αποτελεί κτήμα των τρίτων χωρών. Θα φροντίζουμε να καταπολεμήσουμε την φυγή εγκεφάλων και να ενισχύσουμε τι τις δυνατότητες που δίνονται στους φοιτητές και τους ερευνητές στις χώρες αυτές να βοηθήσουμε ευάλωτες ομάδες, να αντιμετωπίσουμε τις ιδιαίτερες ανάγκες επίσης ε, που έχουν τα άτομα με αναπηρία, μαθησιακές ανάγκες. Πρέπει επίσης να εξασφαλίσουμε ότι θα υποστηριχθεί η συμμετοχή στο πρόγραμμα, το νέο πρόγραμμα Εράσμους ατόμων από, από χώρες με τις οποίες ε, έχουμε αναπτυξιακή συνεργασία. Έτσι ώστε να επιτύχουμε και τους στόχους μας στην, στον τομέα της αναπτυξιακής συνεργασίας. Αγαπητοί συνάδελφοι, όπως πάντοτε προσβλέπω στη συνεργασία που θα έχουμε για να βελτιωθεί το προσχέδιο έκθεσης που σας υποβάλλω. Προσβλέπω στη συζήτηση και μαζί σας και με την κοινωνία των πολιτών, έτσι ώστε να προωθήσουμε τους στόχους μας και στον τομέα αυτών. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Γνάθιο. Θέλει να λάβει το λόγο η Επιτροπή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω αγγλικά. Καλό απόγευμα αγαπητοί συνάδελφοι. Εκπροσωπώ την Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακή Συνεργασία για τα ζητήματα, για τα ζητήματα του λεγόμενου εντίκη. Θα σταθώ σε ορισμένα σημεία. Πρώτα απ' όλα καλωσορίζουμε το προσχέδιο της έκθεσης, νομοδότησης για το πρόγραμμα Εράσμους πράγματι ζητάτε να δοθεί μεγαλύτερη δημοσιότητα, ορατότητα στους, ε, στη διεθνή διάσταση του προγράμματος. Βεβαίω πρέπει να βρούμε τις κατάλληλες διατυπώσει όσον αφορά την εξωτερική δράση για να φαίνεται ότι αυτή η διεθνή διάσταση είναι συμβατή με τις επιδιώξει που έχουμε χρησιμοποιώντας το NDICI. Και γι' αυτό προτείνουμε την εξή δομή. Πρώτα απ' όλα έχουμε το NDICI ως γενικότερο βασικό εργαλείο για την εξωτερική δράση που προωθεί τις αξίες και τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναφέρονται πολλές τέτοιες αξίες, πολλά ζητήματα mainstreaming. Αυτό θα πρέπει να αποτελέσει το γνώμονά μας οποτεδήποτε χρησιμοποιούμε χρηματοδότηση Εράσμου. Η διεθνή διάσταση λοιπόν του προγράμματος Εράσμου προέρχεται από τους στόχους που τίθενται στο NDCI. Οι στόχοι αυτοί κατά την άποψή μας λοιπόν καλύτερα περιγράφονται από το NDICI και τα προγράμματα EPA. Εταιρική σχέση. Από εκεί λοιπόν ξεκινούν οι βασικές αξίες, στόχοι που έχουμε, αναφέρατε ορισμένου από αυτού, την ανάπτυξη των χωρών αυτών, την βοήθεια στι ευάλωτε ομάδες. Ενθαρρύνεται ε, η προσπάθεια να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα αυτά μέσω του NDICI. Θα ήθελα επίσης να σας παραπέμψω στο άρθρο 16, το οποίο αναφέρεται στις χώρες οι οποίες επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα Εράσμους ως συνδεδεμένες χώρες. Πρόκειται για χώρες οι οποίες αποφελούνται και από το NDICI. Ε, για τη σύνδεση αυτών των δύο θα θέλαμε πολύ να δούμε τις ε, προτάσεις σας και τις τροπολογίες που θα υποβάλλετε. Ο Πρόεδρος, σας ευχαριστώ πολύ. Κάποιος άλλος συνάδελφος θα ήθελε να πάρει το λόγο. Κύριε Αντιπρόεδρος. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την γνωμοδότηση. Περιμένω λίγο να βάλετε όλοι τα ακουστικά σας. Λοιπόν, έλεγα ότι καλωσορίζω την, ιδιαίτερα την τροπολογία 2 που αναφέρει πόσο σημαντική ε, είναι η εκπαίδευση, πόσο σημαντικό είναι να έχει κανείς πρόσβαση στις πληροφορίες για τις δυνατότητες που δίνει το πρόγραμμα Εράσμους και επίσης για το γεγονό ότι θα πρέπει να λάβουμε ιδιαίτερη μέρημνα για τις ανάγκες των, ελευ... των ευάλωτων ομάδων. Ότι οι ανάγκες αυτών των ομάδων, όσον αφορά τις μαθησιακές τους ανάγκες δηλαδή, θα πρέπει να λεφθούν ιδιαίτερα υπόψη. Ε, Μιλούμε για άτομα με αναπηρία, μιλούμε για αυτόχθονες πληθυσμούς. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι όλοι αυτοί θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν πλήρως στο πρόγραμμα Εράσμους. Ο πρόεδρος, πριν να δώσω το λόγο στον Ιγνάθιο, θα ήθελα και εγώ να κάνω ένα μικρό σχόλιο. Πιστεύω ότι λίγα είναι τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης που έχουν δημιουργήσει ε, τέτοια συνένεση στους Πολίτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση που απολαμβάνουν τέτοια υποστήριξη από όλου του πολίτε. Είναι ένα πρόγραμμα στο οποίο φαίνεται στην πράξη η αρχή της αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών, μεταξύ της δυνατότητας που δίνεται στους ανθρώπους να έρθουν πιο κοντά και με αυτόν τον τρόπο να αντιληφθούν και την ιδιότητα του πολίτη. Το πρόγραμμα Εράσμου είναι ένα εξαιρετικό πρόγραμμα υπ' αυτή την έννοια και πιστεύω ότι είναι πολύ καλή ιδέα να το επεκτείνουμε και να του δώσουμε και μια διεθνή διάσταση έτσι ώστε να δημιουργήσουμε με στρατηγικό τρόπο αυτές τις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων. Να δημιουργήσουμε ανθρώπινες σχέσεις μεταξύ Ευρωπαίων πολιτών, Ευρωπαίων νέων και νέων σε άλλες περιοχές του κόσμου. θα έλεγα ότι το πρόγραμμα εράσμος είναι το καλύτερο δυνατό εργαλείο που μπορεί να μας εξασφαλίσει αυτές τις σχέσεις. Ας βρούμε με ποιον καλύτερο τρόπο μπορούμε να αξιοποιήσουμε το Erasmus, το NDICI ή οποιοδήποτε άλλο εργαλείο, αλλά ο γενικότερο στόχος θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο συντονισμός έτσι ώστε πραγματικά να ενισχύσουμε τις σχέσεις μεταξύ των νέων. Γιατί είδαμε ότι το πρόγραμμα Εράσμους είναι ένα πρόγραμμα ε, εξαιρετικά μεγάλη στρατηγική σχημασία ε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορούμε λοιπόν να το αξιοποιήσουμε και προ όφελο των γεωστρατηγικών μα επιλογών και αναγκών. Σα ευχαριστώ, συμφωνώ πλήρω μαζί σα. Βλέπετε ότι ο λό... προσπαθώ να μιλήσω ισπανικά. Ο λόγο που μπορώ να μιλήσω ισπανικά είναι επειδή είχα, πάει... είχα συμμετάσχει σε ένα πρόγραμμα Εράσμος πριν 10 χρόνια θα βρεθεί στην Ισπανία. Και πιστεύω ότι τα, από όλες τις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το πρόγραμμα Εράσμους ήταν ένα από, το, τα καλύτερα αποτελέσματα που είχε. Και αν μπορέσουμε τελικά να συμπεριλάβουμε σε αυτό και παιδιά και νέους από τις αναπτυσσόμενες χώρες, αυτό είναι θα ήταν εξαιρετικό και για μας και για το μέλλον αυτών των παιδιών και για το μέλλον αυτών των χωρών. Έρχομαι τώρα στην τροπολογία υπεριθμών 2. Βεβαίως υποστηρίζουμε την πρότασή σας να συμπεριλάβουμε και τους αυτόχθονες πληθυσμούς. Ε, μπορούμε, αν το υποβάλλετε, να το συμπεριλάβουμε και στο κείμενο. Συμφωνούμε επί της ουσίας πάντως 100% και Διαπιστώνω επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι ο NDCI είναι το καλύτερο εργαλείο. Αμφιβάλλουμε όμως εμείς θεωρούμε ότι ίσως υπάρχουν κάποια δομικά προβλήματα στον τρόπο με τον οποίο είναι φτιαγμένο, στημένο το NDCI. αμφιβάλλουμε για το αν ε, το εργαλείο τελικά θα λειτουργήσει ακριβώς όπως περιγράψετε. Θα δούμε. Ευχαριστώ. Στη... Στη Γαλλικία είχατε, είμαι σίγουρος, περάσει το πρόγραμμα Erasmus σας. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι δεν έχουμε πολύ χρόνο εξαιτίας του χρονοδιαγράμματος της ε, καθήλυνα αρμόδια επιτροπή Κουλτ για να παρουσιάσουμε τις τροπολογίες. Η προθεσμία είναι 22 Νοεμβρίου, δηλαδή 10 το πρωί, δηλαδή αυτή την Πέμπτη 10 το πρωί. Και θα οργανωθεί και έκτακτη ε, συνάντηση στο Στρασβούργο είτε στις 10 είτε στις 13 ε, Δεκεμβρίου. Χρειάζεται να περιμένουμε ή μπορούμε να συνεχίσουμε το επόμενο σημείο της μέρη τη διάταξης, ρωτά ο Πρόεδρος. Ένα μικρό διάλειμμα χρειάζεται. María. Thank you. Gracias. Ο πρόεδρος λέει ευχαριστώ σε διάφορες γλώσσες. Σου δίνω και λίγο χρόνο να βάλεις τα ακουστικά σου. Αν τα πούμε στα αγγλικά ώστε να μην χρειάζεται μετάφραση από τα ισπανικά. Νομοθετική πρόταση για τα τρία σχέδια κανονισμών της Επιτροπής, δηλαδή κοινή αγροτική πολιτική στρατηγικό σχέδιο, οριζόντιος κανονισμός και τροποποιητικός κανονισμός που συναποτελούν μέρη του ίδιου νομοθετικού πακέτου με στόχο να αναθεωρηθεί η τρέχουσα ΚΑΠ. Οι στρατηγικοί κανονισμοί καλύπτουν άμεσες πληρωμές, άμεσες καταβολές στους γεωργούς, ανάπτυξη υπαίθρου και τομεακά προγράμματα στήριξης. Ο οριζόντιος κανονισμός ΚΑΠ καλύπτει τη χρηματοδότηση και παρακολούθηση της ΚΑΠ. Και ο τροποποιητικός ε, κανονισμός για την ενιαία οργάνωση αγορών για ποιοτικά προγράμματα αγροτικών προϊόντων και ειδικά μέτρα για υπερπόντιες περιοχές και μικρά νησιά του Αιγαίου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την πρότασή της πρώτη η του 18 και περιγράφει πώς προτίθεται να αναθεωρήσει την κοινή αγροτική πολιτική πέραν του 2021. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021 έως 2027 περιλαμβάνει 365 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία αντιστοιχούν σε 28,5% του συνολικού κοινοτικού προϋπολογισμού για την περίοδο 2021 έως 2027. Από το ποσό αυτό, 265,2 δισεκατομμύρια προβλέπονται για άμεσες καταβολές, 20 δισεκατομμύρια για μέτρα στήριξης αγοράς και 78,8 δισεκατομμύρια για την ανάπτυξη πέθρου με τη νέα κοινή αγροτική πολιτική. Η Κομισιόν στοχεύει σε βελτίωση της ανταπόκρισης στις νέες οικονομικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις, στην ευθυγράμμιση των στόχων με τις 10 προτεραιότητες του Πρόεδρου Γιούνκερ και, τις, και τους στόχους μάλλον βιώσιμης ανάπτυξης και την απλούστευση της εφαρμογής. Έχει και σχέδια για περισσότερο για μια προσέγγιση περισσότερο βασισμένη στην απόδοση και να δώσει περισσότερο λόγο σε μεγάλε χώρε μέλη στη διαμόρφωση τη κοινή αγροτική πολιτική. Το Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα με τίτλο Το μέλλον τη διατροφή και τη αγροτική καλλιέργεια στι 30 Μαου 2018, πριν από την επίσημη παρουσίαση της, ε, των προτάσεων κοινή αγροτική πολιτική. Ο στόχο του ήταν να διαμορφώσει τι τρει νομοθετικές προτάσεις, αλλά βέβαια επέτυχε εν μέρη μόνο. Η συγγήτριά μας για τις γνωμοδοτήσεις είναι η κυρία Χόιμπουχ, στην οποία τώρα παραδίδω τον λόγο. Ως γνωρίζουμε, η Μαρία είναι πραγματική ειδήμων στον τομέα της αγροτικής οικονομίας. Άλλωστε συνεργαστήκαμε και μαζί μου, λέει ο κ. Γκερέρο, σε συνάντηση του ΦΑΟ στη Μαδρίτη σχετικά με την ασφάλεια ε, διατροφής δηλαδή και άλλων σχετικών θεμάτων και άλλα σχετικά θέματα μάλλον και τα τελευταία πέντε χρόνια έχουμε κατ' επανάληψη δει και θαυμάσει την εμπειρογνωμοσύνη σου στα θέματα αυτά. Ευχαριστώ πολύ, Ενρίκε. Όμω θα συνεχίσω στα γερμανικά. Φορέστε αμέσω τα ακουστικά σα για να καταλάβετε τι θα λέω. Αγαπητέ και αγαπητοί συνάδελφοι, μάλλον αγαπητοί συνάδελφοι, γιατί σας δεν βλέπω, είχατε χρόνο για να κοιτάξετε τις γνωμοδοτήσεις, τα σχέδια δηλαδή, θα είδατε ότι δεν περιλαμβάνουν πολλά νέα στοιχεία, άλλωστε αυτά τα έχουμε ξαναπεί τα περισσότερα και πράγματι στην γνωμοδότησή μου επαναλαμβάνονται γνωστές απαντήσεις σε ένα παλαιό πρόβλημα, δηλαδή στην έλλειψη συνοχής της κοινή αγροτικής πολιτικής της Ευρώπης, έλλειψη συνοχής με τους στόχους της αναπτυξιακής συνεργασίας. Η Επιτροπή μας έχει εγγύψει ε, σοβαρά στο θέμα αυτό στην παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο. Θα θυμάστε και την κοινή μας συνεδρίαση την Άνοιξη με την Επιτροπή Γεωργίας και τα, με, τα αποτελέσματα μελέτης την οποία αναθέσαμε ως κοινοβουλευτική επιτροπή που συζητούσαμε τις καταστροφικές συνέπειες της εξαγωγής γαλακτοκομικών στην Αφρική για ντάμπινγκ στον τομέα των πουλερικών, για την αγροτική βιομηχανία στην Ευρώπη η οποία εξακολουθεί να υπερθερμαίνει το κλίμα, αλλά και στην προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο η Επιτροπή Αναπτυξιακής Συνεργασίας είχε ασχοληθεί με την κοινή αγροτική πολιτική. Όταν άρχισα την εργασία μου επί της γνωμοδοτήσεως, επέλεξα τα σημεία εκείνα τα οποία η Επιτροπή μας είχε ήδη εγκρίνει το 2011. Το 2011 λοιπόν η τότε εισηγήτρια του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή ΔΕΒΕ και στην γνωμοδότησή της ε, ήταν μια συνάδελφός μας Γερμανίδα από το Τσέντεου άρχιζε με την εξής φράση την οποία θα σας διαβάσω τώρα. Τι έλεγε τότε λοιπόν. Από την οπτική της αναπτυξιακής πολιτικής θα έπρεπε να διαμορφωθεί μια πολύ διαφορετική κοινή αγροτική πολιτική από αυτήν που διαλαμβάνει η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτά έλεγε τότε η συνάδελφός μας. Και σήμερα εγώ δεν μπορώ παρά να επαναλάβω την φράση αυτή. Η γνωμοδότης του 2011 προτείνει πλέον σημαντικά μέτρα ώστε να αντιμετωπιστούν οι αρνητικές επιπτώσεις της κοινή αγροτικής πολιτικής ή τουλάχιστον να μετριαστούν. Οι προτάσεις αυτές, επαναλαμβάνω το 2011, επανέρχονται στην γνωμοδότησή μου. Τις επαναλαμβάνω, διότι εξακολουθούν να είναι επίκαιρε και ισχυρές. Σε σύγκριση με το 2011, τονίζω εγώ στην γνωμοδότησή μου επίσης το θέμα του κλίματος, που είναι πια πάρα πολύ ε, έντονο και μετά μάλιστα από το πολύ θερμό καλοκαίρι που περάσαμε και προβάλλω και σε νέες τεχνικές τροπολογίες, περισσότερες πολιτικές απαιτήσει, διότι δεν αρκεί να μιλήσουμε μόνο για την αναπτυξιακή συνεργασία και να περιλαμβάνουμε κάποιους στόχους στο αιτιολογικό της ε, προτάσεως, δηλαδή στα εκτιμώντας, πρέπει να μπουν στο διατακτικό και να λάβουν συγκεκριμένη μορφή. Να μου επιτρέψετε τώρα, μάλλον θα με ρωτήσετε, καλή ήταν η γνώμοδος 2011 και σε αυτήν μπορεί κανείς να βασιστεί. Όμως, δεν σημαίνει αυτό ότι οι προτάσεις που έγιναν τότε στη γνωμοδότηση τελικώς δεν τηρήθηκαν, δεν ελήφθηκαν υπόψη. Σωστό είναι αυτό. Πράγματι, η Επιτροπή Γεωργίας δεν υιοθέτησε τις καλές αυτές προτάσεις της γνωμοδοτήσεως μας, της Επιτροπής μας δηλαδή του 2011. Παρ' όλα αυτά, εγώ ελπίζω ότι θα έχουμε τώρα μεγαλύτερη επιτυχία. Ελπίζω τα πράγματα να πάνε διαφορετικά, διότι από το 2011 πολλά έχουν γίνει. Το 2015 ζήσαμε την κρίση του μεταναστευτικού, η οποία ε, επέσυρε την προσοχή μας στα θέματα αυτά και στην έλλειψη συνοχής της πολιτικής και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και εκτός αυτού, δηλαδή ε, στο κοινό. Ο δε νυν Επίτροπος Γεωργίας Χόγκαν ίδρυσε και ειδική task force για την Αφρική. Δηλαδή και από την πλευρά της πολιτικής για την γεωργία αντιλαμβάνονται πλέον ότι υπάρχουν προβλήματα και ιδίω για και στην Αφρική. Αυτή η Task Force επεξεργάζεται τώρα συστάσεις και για τούτην εδώ την αναθεώρηση. Και αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για μας. Στην ανακοίνωση δε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που προηγήθηκαν της νομοθετικής προτάσεως περιλαμβάνεται και ιδιαίτερο κεφάλαιο για την ανάπτυξη. Με λίγα λόγια, Έχουμε τώρα μια διαφορετική αφετηρία από αυτήν του 2011. Έχουμε λοιπόν τώρα μια όρμη, ένα momentum που θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε πολιτικά. Θα έλθω στα πιο σημαντικά ουσιώδη θέματα των τριών σχεδίων μου γνωμοδοτήσεων. Μιλούμε για τρεις γνωμοδοτήσεις όπως είπε και ο Προεδρεύων πριν, διότι έχει τρία σκέλη νομοθετική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δηλαδή τρεις διαφορετικούς κανονισμούς. Πυρήνας του κανονισμού ή των κανονισμών είναι τα στρατηγικά σχέδια. Μάλλον ο κανονισμός για το στρατηγικό σχεδιασμό. Ο κανονισμός αυτός διατυπώνει στόχους της κοινή αγροτικής πολιτικής, δηλαδή τι θα πρέπει να επιτευχθεί. Διατυπώνει επίσης τα μέσα ή τα όργανα, δηλαδή το πώς θα επιτευχθούν οι στόχοι. Αναφέρεται και στους τομείς και ποιες μέθοδοι παραγωγής ή ποιοι τρόποι παραγωγής θα πρέπει τελικώς να στηριχθούν. Ο κανονισμός αυτός είναι σημαντικός από την άποψη της πολιτικής συνοχής για την ανάπτυξη. Με την υποστήριξή σας επιθυμώ να τροποποιήσω τις εξής έξι πτυχές του κανονισμού αυτού. Πρώτο, θα πρέπει να περιλαμβάνεται ρητή δέσμευση υπέρ της συνοχής της πολιτικής. Διότι κάτι τέτοιο δεν υπάρχει στο τμήμα περιστόχων και ακριβώς εκεί πρέπει να μπει αυτή η δέσμευση. Τις, σημαντικές, τις, σημαντικές, τις σημαντικότερες τροπολογίες θα βρείτε ως, με αριθμούς 4, 24 και 36. Δεύτερο, σύντομο κεφάλαιο για την ανάπτυξη, το οποίο να ξεκαθαρίζει ότι η κοινή αγροτική πολιτική εξυπηρετεί στην προσπάθεια επίτευξη των στόχων SDG, δηλαδή βιώσιμης ανάπτυξης. Διότι για την ώρα η διάσταση της αναπτυξιακής πολιτικής δεν είναι ορατή στον κανονισμό. Οι πιο σημαντικές τροπολογίες είναι 39, 40 και 41. Τρίτο, χρειαζόμαστε συστηματικό monitoring των επιπτώσεων της κοινή αγροτικής πολιτικής στην αναπτυξιακή συνεργασία. Διότι για την ώρα, παρόλο που θα ήταν μεθοδολογικά δυνατό, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν συλλέγει σχετικά δεδομένα. Και εδώ αναφέρουμε στις τροπολογίες 62-67. Τέταρτο, πρέπει να εξασφαλιστεί ότι οι επιδοτήσεις, και εδώ αναφέρομαι ιδίω στις συνδεδεμένες πληρωμές, δεν θα προκαλούν ζημία, διότι για την ώρα οι συνδεδεμένες αυτές πληρωμέ έχουν και αρνητικέ επιπτώσει, ιδίω στον τομέα τη ζάχαρη. Για αύριο προβλέπεται μάλιστα και συζήτηση με εταίρου των, των χωρών ΑΚΕ. Γνωρίζουμε λοιπόν το πρόβλημα και γι' αυτό εγώ προτείνω ένα σύνολο κριτηρίων που θα πρέπει να πληρούνται όταν χώρες μέλη καταβάλουν συνδεδεμένες πωλήσει για ένα συγκεκριμένο προϊόν. Οι τροπολογίες μου είναι 12, 16, 46 48 και 49. Πέμπτο, η επέκταση της υποστήριξης για λευκοματούχα φυτά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να μειωθεί η εξάρτησή μας από εισαγωγές σόγιας. Για την ώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι σε θέση να αυξήσει τις πρωτεΐνες που είναι αναγκαίες για διατροφή των ζώων και μεταφέρει τεράστιες ποσότητες σόγιας από την Νότια Αμερική. Και δεν μιλούμε για οποιαδήποτε σόγια, μιλούμε για σόγια η οποία είναι γενετικά τροποποιημένη, προέρχεται από μονοκαλλιέργειες, από φτωχού αγρότες και αγρότησες που εργάζονται υπό δεινές συνθήκες εργασίας. Πρέπει με την αναθεώρηση της ΚΑΠ η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει την ευθύνη για το σύνολο της αλυσίδας προμήθειας. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν όχι μόνο εμείς να γίνουμε αυτάρκης σε πρωτεΐνες, αλλά να διαφορούμε και τις συνθήκες υπό τις οποίες ε, καλλιεργούνται τα, πρωτο, τα πρωτεϊνούχα φυτά. Και εδώ είναι η τροπολογία 50 Χρειαζόμαστε καθορισμό ελάχιστων ε, προδιαγραφών για το περιβάλλον που να είναι υποχρεωτικά δεσμευτικές για τις πληρωμές που θα γίνονται ώστε να αντιμετωπιστούν οι αρνητικέ, οικολογικές και κλιματικές συνέπειες ή τουλάχιστον να μετριαστούν. Είναι πραγματικό, πραγματικός φωνιάς του κλίματος η αγροτική παραγωγή με 11% συμμετοχή στην εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου. Και γνωρίζουμε πολύ καλά ποιες είναι οι τρομερές συνέπειες των ε, ε, καταστροφών που έρχονται από την αλλαγή του κλίματος η συνοχή της πολιτικής πρέπει να, λάβει, μάλλον, πρέπει να θεωρήσει το κλίμα ύψιστη προτεραιότητα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και δεν επιτρέπεται σε ό,τι αφορά τις ειδήσει που έρχονται για το κλίμα να τις αντιμετωπίσει με ενοχελικό τρόπο. Γι' αυτό έχουμε και πολλές τροπολογίες εδώ, 38, 44, 45 και 47 διότι οι συνέπειες της αλλαγής του κλίματος πλήττουν και τους Ευρωπαίους γεωργούς και αγρότες και αγρότησες, αλλά βεβαίως και τους ομολόγους τους σε όλο το νότιο ημισφαίριο. Τώρα, αν με αφήσει βέβαια η φωνή μου που αρχίζω να τη χάνω σιγά σιγά, για τον οριζόντιο κανονισμό λίγα πράγματα, τα όσα είπα μόλις αναφέρονται και σε τον εδώ τον κανονισμό, όχι μόνο τον κανονισμό για τον στρατηγικό σχεδιασμό, πρέπει και στον οριζόντιο κανονισμό να εξετάσουμε και να ορίσουμε τα πράγματα με μεγάλη ακρίβεια. Πρόκειται για τους κανόνες της χρηματοδότησης. Και εδώ λοιπόν πρέπει να εξηγήσουμε ακριβώς τι θέλουμε. Πρόκειται για το management, πρόκειται για το monitoring, μέσα στα πλαίσια της αναθεώρησης της ΚΑΠ. Εγώ προτείνω εδώ διάφορες τροπολογίες, οι οποίες απορρέουν από αυτές που ανέφερα προηγουμένως, ώστε να κινούμαστε παραλλήλως προς την ίδια κατεύθυνση. Οι σημαντικότερες τροποποίησεις είναι η διεύρυνση του συστηματικού monitoring, είναι οι διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμφεροντούχους δηλαδή των χωρών εταίρων, πρόκειται για τις δημοσιονομικές συνέπειες για τις χώρες μέλη όταν δεν τηρούν τις αρχές της πολιτικής συνοχής και εδώ χρειαζόμαστε λοιπόν κάποιο μέσον πίεσης και λίγα λόγια τώρα για τον τρίτο κανονισμό, που είναι και ο τελευταίος και που είναι η κοινή οργάνωση αγοράς και που διευκρινίζει ποιες παρεμβάσεις γίνονται στις αγορές, ποιες βοήθειες, ποια μέτρα α, κατεπήγοντος λαμβάνονται ή επιτρέπεται να λαμβάνονται και εδώ οι τροπολογίε μου περιορίζονται ιδίω σε ένα γνωστό πρόβλημα. Δηλαδή έχουμε υπερπαραγωγή στην Ευρώπη που οδηγεί βεβαίως σε φτηνές εξαγωγές αγροτικών προϊόντων. Το καλύτερο παράδειγμα είναι η σκόνη γάλακτος. Έχουμε ακόμα στις αποθήκες 90.000 τόνους γάλακτος σε σκόνη από την τελευταία κρίση και αντί να προσαρμόσουμε την παραγωγή στις ανάγκες της αγοράς έχουμε κάνει και παρεμβάσεις. Εγώ προτείνω ένα πρόγραμμα για την εθελοντική μείωση των παραγωμένων ποσοτήτων είναι τελικώς πιο οικονομικό να παράγεται λιγότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρά να γίνονται παρεμβάσεις και μετά να πετάγεται αυτό, να γίνεται dumping δηλαδή σε άλλες αγορές όπου βεβαίως δεν ε, ωφελούνται οι γαλακτοπαραγωγοί στην Ευρώπη. Είναι άλλωστε προφανές ότι η πίεση επί της αγοράς εξακολουθεί. Εδώ στην Ευρώπη η τιμή του γάλακτος δεν έχει ανέβει και όπως είπα υπάρχουν και 90.000 τόνοι στις αποθήκες. Αξιότιμες και αξιότιμοι συνάδελφοι, λοιπόν, αυτά είναι τα πιο σημαντικά από τα σχέδια που έχω υποβάλει για τις τρεις γνωμοδοτήσεις και με μεγάλη χαρά θα συζητήσω τώρα μαζί σας και θα ακούσω τις προτάσεις σας. Ευχαριστούμε πολύ Μαρία. Πριν προχωρήσουμε θα ήθελα να καλωσορίσω τον κύριο Πόγκα ο οποίος δεν είχε έρθει εδώ και καιρό στο Κοινοβούλιο. Έρχεται από πολύ μακριά. Πάντα τον αισθανόμασταν κοντά, βέβαια. Συγχαρητήρια λοιπόν για το νυν κοινοβουλευτικό σας έργο. Ο κύριος Στέφαν Κέρολτ έχει το λόγο ως κοιόδης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και εσάς κύριε Συγήτρια, κυρίες και κύριοι. Θέλω πρώτα να ευχαριστήσω, ξαναλέω, την εισηγήτρια για τα σχέδιά της. Στο παρελθόν, οι ενδεχόμενες επιπτώσεις της κοινή αγροτικής πολιτικής στις αναπτυσσόμενες χώρες δεν λαμβάνονταν πάντοτε υπόψη. Αυτό το έφτιαξε ήδη η εισηγήτρια. Τα σχέδια που έχει υποβάλει δείχνουν σε ποιο βαθμό μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ευκαιρία τη αναθεώρησης τη κοινή αγροτική πολιτικής ώστε να βελτιωθεί η συνοχή της πολιτικής υπέρ των αναπτυσσόμενων χώρων. Συμφωνώ με πολλού από τους διατυπωμένους στόχους. Βέβαια, στο πώς θα επιτευχθούν οι στόχοι υπάρχουν διαφορετικές αντιλήψεις. Και εγώ λοιπόν με τη σειρά μου θα καταθέσω τροπολογίε. Έχω περάσει αρκετά χρόνια τη ζωή μου στην Σαχέλ, και έχω ιδιαίτερο ενδιαφέρον για θέματα ε, ανάπτυξης και γι' αυτό είμαι και αναπληρωματικό μέλος εδώ παροιμήν. Με ενδιαφέρει τώρα η συνεργασία, η κοινωνική πολιτική στα πλαίσια της συνεργασίας και πρέπει να λαμβάνετε υπόψη και, και θα πρέπει να λάβουμε και σοβαρά υπόψη την εντολή που δίνουν οι συνθήκες για την ένταξη όλων των χωρών στην παγκόσμια οικονομία. Αυτό σημαίνει και σταδιακή μείωση των ε, φραγμών στο εμπόριο, συμπόρευση οικονομικής και αγροτικής πολιτικής που θα ωφελήσει όλους και βεβαίως και τις αναπτυσσόμενες χώρες. Λαμβάνοντας υπόψη την κοινή μας ευθύνη απέναντι πρώτα στην προσπάθεια απάλληψη της φτώχειας, δεύτερο στην βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος, τρίτο στην βιώσιμη ανάπτυξη των απανταχού φυσικών πόρων. Θα πρέπει να βρούμε τρόπο να διατηρήσουμε τις ελευθερίες μας, να τις προωθήσουμε και εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπέρ των παραγωγών αλλά και υπέρ των καταναλωτών έχω την εντύπωση ότι ορισμένες από τις προτάσεις που, καν, που γίνονται στην, στα σχέδια γνωμοδοτήσεων δεν λαμβάνουν επαρκώς υπόψη τις ελευθερίες αυτές. Υπάρχει όμως η δυνατότητα να δοθούν κίνητρα σε επιχειρήσεις και να οδηγηθούν έτσι σε συνεργασίες με αναπτυσσόμενες χώρες που να προωθήσουν την ανάπτυξη. Το γεγονό ότι οι μηχανισμοί της κοινή αγροτικής πολιτικής έχουν ενδεχομένως επιπτώσεις σε αναπτυσσόμενες χώρες, πρέπει να μετρηθούν σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματά τους. Θα πρέπει να είναι δυνατόν να επιτευχθεί η ευρύτερη δυνατή συνένεση και να δοθεί ένα ξεκάθαρο μήνυμα, διότι μόνον έτσι μπορούμε να αναμένουμε ότι η γνωμοδότησή μας θα ληφθεί επαρκώς υπόψη και ότι οι νομοθετικές προσπάθειες θα αποδώσουν καρπούς. Αναμένω με ενδιαφέρον γόνιμη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή συγγνώμη, με την εισηγήτρια, αλλά και με τους σκιώδεις και τις σκιώδεις εισηγήτριες και άλλα μέλη της Επιτροπής Αναπτύξεως. Θα πρέπει να βρούμε μια ισορροπία ανάμεσα στην προστασία των παραγωγών μας, διατήρηση της ανταγωνιστικότητας και σεβασμό των διεθνών μας υποχρεώσεων στον τομέα της αναπτύξεως. Σας ευχαριστώ πολύ. Maria. Kiitoksia Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω και πάλι στα φινλανδικά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια. για την παρουσίαση που μας έκανε για τις ε, γνωμοδοτήσεις, τη γνωμοδότησή της. Συχνά συμφωνούμε. Ωστόσο θα ήθελα να σταθώ σε τρία θέματα. Πρώτον, Συμφωνώ και εγώ ότι πρέπει να είναι πρώτη μας προτεραιότητα η προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης μέσω της ΚΑΠ. η πρόθεση της βιώσιμης ανάπτυξης συνδέεται και με την αναπτυξιακή συνεργασία. Συχνά συζητούμε για θέματα όπως για παράδειγμα η μέθοδη παραγωγής, η ποιότητα του εδάφους, που βλέπουμε τη σύνδεση με την οποία υπάρχει. Έτσι ώστε η γεωργία να προσαρμοστεί, να σέβεται το περιβάλλον, να ε, μην δημιουργεί προβλήματα με την ποιότητα του εδάφους ή άλλα. Προστασία λοιπόν του περιβάλλοντος κατά την άποψή μου θα πρέπει να βρίσκεται στο κέντρο της ε, πρότασής μας. Δεύτερον, έχουμε αυτό το αιώνιο ε, ερώτημα συζήτησης, ε, θέμα συζήτησης ε, της στόχευσης των ενισχύσεων. Όμως εμείς πρέπει να δούμε το ζήτημα από την πλευρά της Επιτροπής ΔΕΒΕ, την πλευρά της αναπτυξιακής συνεργασίας δηλαδή, και να πούμε ότι το σημαντικό θα είναι οι ενισχύσεις να οδηγούν σε βελτίωση της τοπικής παραγωγής του, του των μικρών παραγωγών επιτόπου. Τρίτο θέμα. Εσυγήτρια αναφερθήκατε στο γεγονό ότι υπάρχει υπερπαραγωγή τροφίμων, ορισμένων τροφίμων και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε ορισμένες περιπτώσεις και σε παγκόσμιο επίπεδο. Αναφερθήκατε για παράδειγμα για το γάλα σε σκόνη. Και η λύση που προτείνατε ήταν η μείωση της παραγωγής. Όμως τι ακριβώς εννοείτε, πώς θα γινόταν αυτό με οικονομικά κίνητρα, πώς. Θα, θα ήθελα να μου απαντήσετε σε αυτές τις τρεις ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελε κάποιος άλλος συνάδελφος το λόγο. Η Επιτροπή. Μία. Λε, ονομάζεστε, παρακαλώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Το πολλά θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για τα προσχέδια γνωμοδοτήσεων που μας παρουσιάζει και τις πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις που είχαμε, που έχουμε. Χωρισμένα συγκεκριμένα σχόλια, παρατηρήσεις για τις τροπολογίες Προηγουμένω όμως θα ήθελα να υπενθυμίσω ποιο είναι ο στόχος της αναθεώρησης της ΚΑΠ και τι επιδιώκουμε. Το οποίο συνδέεται με κάτι που ανέφερε και η αντιπρόεδρό σα για το ζήτημα τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η βιώσιμη ανάπτυξη βρισκόταν στο κέντρο τη διαδικασία αναθεώρηση τη ΚΑΠ, η οποία δεν ξεκίνησε τον Ιούνιο, αρχέ Ιουνίου, όταν υποβάλαμε τι προσπάθειέ μα, αλλά πολύ νωρίτερα, ήδη από το 2017, όταν ξεκινήσαμε τι διαδικασίε διαβούλευση, όταν έγιναν οι σχετικέ ανακοινώσει τη Επιτροπή, στι οποίε επανειλημμένα αναφερθήκαμε στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και στο πόσο σημαντικό είναι η ΚΑΠ να ε, προωθεί τους στόχους προστασίας του περιβάλλοντος συμπεριλαμβανομένων και των στόχων που έχουμε θέσει για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και την επίτευξη της Συμφωνίας των Περαισίων. Αυτό μεταφράζεται και στα εργαλεία τα οποία προτείνουμε, αλλά επίσης και στον τρόπο με τον οποίο θα καταρτίζεται η πολιτική αυτή στο μέλλον έτσι ώστε να συνεισφέρουμε στους στόχους αυτούς. Για πρώτη φορά εγκαταλείπουμε το λεγόμενο σύστημα συμμόρφωσης, με το οποίο ουσιαστικά η Ευρωπαϊκή Ένωση περιέγραφε πολύ αναλυτικά τι θα ε, έπρεπε να κάνει κανείς, ε, τους πολιτικούς στόχους και τον τρόπο επιτευξής τους. Το νέο σύστημά μας έχει, ε, βασίζεται στις επιδόσεις. Καταρτίζουμε εννέα βασικούς στόχους, και μετά τα κράτη-μέλη έχουν την ελευθερία να ε, λάβουν υπόψη τους τις εθνικές τους ιδιωτερότητες και τις εθνικές τους ανάγκες και να αποφασίσουν πώς θα τους επιτύχουν αυτούς τους στόχους. Το έχουμε αντιληφθεί ε, το είχαμε αντιληφθεί και με την Ευρώπη των 28 και τώρα με την Ευρώπη των 27, ότι δεν είναι δυνατόν το ίδιο μοντέλο να εφαρμοστεί σε όλους one size fits all. Χρειάζεται να λαμβάνονται υπόψη οι τοπικές ιδιαιτερότητες. Τρει από αυτού τους στόχου αναφέρονται συγκεκριμένα στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγή και την προστασία του περιβάλλοντος. Και προτείνουν μια σειρά εργαλείων από, από τα οποία μπορούν να επιλέξουν τα κράτη-μέλη αυτά που προτιμούν Πρώτα απ' όλα υπάρχει μια, ένα νέο σύστημα αιρεσιμότητας, αξιοποιώντας τις εμπειρίες που είχαμε από το greening, από το πρόγραμμα οικολογικοποίησης και όσον αφορά τον πρώτο πυλώνα, αλλά και όσον αφορά ορισμένες earmarked ξεχωριστές χρηματοδοτήσεις του δευτέρου πυλώνα. Όμως κατά την άποψή μου το σημαντικό είναι ότι οποτεδήποτε πλέον τα κράτη-μέλη θα έρχονται, θα απευθύνονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα υποβάλουν τα σχέδιά τους, θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι με τα σχέδια τους αυτά βελτιώνεται η προστασία του περιβάλλοντος, βελτιώνεται η επίτευξη των, της βιώσιμης ανάπτυξης. Θα πρέπει να φαίνεται λοιπόν ότι τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα αξιοποιούνται προς την κατεύθυνση αυτή. με τις τροπολογίες συμφωνούμε επί της ουσίας, συμφωνούμε με αυτό που επιδιώκεται, όμως ίσως έχουμε μια διαφορετική προσέγγιση στο πώς θα επιτευχθεί. Σας μίλησα για μια, ε, ένα μενού, μια παλέτα με ε, εργαλείων, το οποίο καταγράφεται στο παράρτημα 11 και το οποίο μπορούν, από τα οποία μπορούν να επιλέξουν τα κράτη-μέλη όταν καταπτύσσουν τις στρατηγικές τους. θα βρείτε εκεί και απαντήσεις σε άλλα θέματα που αναφέρατε, όπως για παράδειγμα τη διαχείριση της αγοράς, των εξελίξεων στην αγορά. Η εισηγήτρια ανέφερε ότι πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε προσανατολισμένοι στη διαχείριση των, της αγοράς. Το είναι σημαντικό όχι μόνο στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά επίσης και σε εξωτερικό επίπεδο. είναι πολύ καλύτερο να έχει κανεί μια προσέγγιση που να βασίζεται στην αγορά για να επιτύχει τρόφιμα τα οποία να ανταποκρίνονται στι ανάγκε του. Ε, πολύ περισσότερο από ότι να προσπαθήσει ένας νομοθέτης να περιγράψει αναλυτικά όλους τους κανόνες. Έχουμε συγκεκριμένα μέτρα για ορισμένα ε, γεωργικά προϊόντα, ε, το, το νίνο, το γάλα, ε, την ζάχαρη, είχαμε σχετικές εμπειρίες δηλαδή στο παρελθόν. Και ε, Αυτός πρώτο σχόλιο. Μιλήσατε επίσης για το ζήτημα των συνδεδεμένων ενισχύσεων. Ε, νομίζω ότι έχουμε λάβει υπόψη μας ε, επαρκώς τα προβλήματα ή τις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν αυτές οι συνδεδεμένες ενισχύσεις και έχουμε θέσει προϋποθέσεις. Δηλαδή, τα κράτη-μέλη μπορούν να αξιοποιούν τις συνδεδεμένες ενισχύσεις μόνο όταν πρόκειται για έναν κλάδο ο οποίος βρίσκεται σε οικονομική δυσπραγία ε, με, με, με, και υπάρχει και συγκεκριμένη ποσόστοση που περιορίζει την χρήση τους. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ε, ε, επίπεδο ελέγχου, είναι το επίπεδο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε εμάς θα υποβάλλουν τα στρατηγικά του σχέδια τα κράτη-μέλη, θα δούμε τις συνδεδεμένες ενισχύσεις που προτείνουν και αν θεωρήσουμε ότι ε, υπερβάλλουν, θα τους υποβάλουμε ερωτήματα. Αναφερθήκατε επίση και για το ζήτημα των πρωτοεινούχων φυτών. Τι επόμενε εβδομάδε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει μια ένα πρόγραμμα το οποίο συνοψίζει και τις πολλές πρωτοβουλίες που ήδη είχαν αναλάβει τα κράτη-μέλη για να υποστηρίξουν αυτόν τον κλάδο. Ε, υπάρχει μια ιδέα για μια επιπλέον ενίσχυση πέραν του 10% της συνδεδεμένης ενίσχυσης, ειδικά για τις καλλιέργειες πρωτοενούχων φυτών. Θα έλεγα λοιπόν ότι συνολικά στι προτάσεις μας θα μπορέσετε να βρείτε διάφορα στοιχεία που ανταποκρίνονται στι επιδιώξει σα. Θα δούμε πώ θα συνεργαστούμε και με τη δική σα επιτροπή και με τι άλλε επιτροπέ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έτσι ώστε να καταλήξουμε σε ένα τελικό κείμενο που να ανταποκρίνεται στις επιδιώξει όλων. Υπό αυτή την έννοια προσβλέπουμε στον τριμερή διάλογο μαζί σα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Η Μαρία έχει το λόγο και πάλι. Ευχαριστώ πολύ αγαπητή Πρόεδρε. Από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είπατε πολλά θεμελιώδη πράγματα για την αναθεώρηση της ε, αγροτικής πολιτικής. Δεν χρειάζεται βέβαια να τα συζητήσουμε τώρα. Αυτά θα συζητηθούν στην Γεωργική Επιτροπή όπου σίγουρα θα συμμετέχετε για τον ε, βασικό προσανατολισμό δηλαδή. Τονίσατε και πάλι ότι η βιωσιμότητα βρίσκεται στο επίκεντρο. Και εγώ νομίζω ότι αυτά συνδέονται πολύ στενά μεταξύ τους. Για το μέλλον θα πρέπει να κινηθούμε με πολύ πιο βιώσιμο τρόπο. Αυτή είναι και η πρόθεσή μου με τις τροπολογίες που καταθέτω. Η βιωσιμότητα δηλαδή να μην μείνει μονάχα μια κοινή κουβέντα, αλλά να μπει πραγματικά στα θεμέλια. Είμαι διαθέσιμη να συνεργαστώ μαζί σας ε, επικοδομητικά. Νομίζω ότι τα συμφέροντά μας, τα ενδιαφέροντά μας αν θέλετε καλύτερα, ε, κινούνται προ την ίδια κατεύθυνση. Και θα ε, συμβάλλω στην προσπάθεια αυτή με τι τροπολογίε μου. Τώρα για τις συνδεδεμένε πληρωμές, γιατί και αναφέρθηκα σε αυτέ προηγουμένω, χαίρομαι που τις περιορίζετε στο 10%. και τη συνδέεται με συγκεκριμένους όρους. Και εδώ μπορούμε να ενισχύσουμε την πορεία αυτή. Εάν οι συνδεδεμένες πληρωμές δεν ζημιώνουν την αγορά, αν έχουν σημαντική ωφέλεια για το περιβάλλον, τότε νομίζω ότι πράγματι μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως κατάλληλο μέσο. Αν πούμε όμως απλώς, να, για το κρέας ή για το γάλα κάνουμε συνδεδεμένες ε, πληρωμές ε, έτσι κατά το δοκούν, αυτό δεν έχει κανένα νόημα, το έχουμε δει και έχουν οδηγήσει και σε ε, επιζήμιες συνέπειες στο παρελθόν. Τελευταία φράση για την υπερπαραγωγή και πώς θα περιοριστεί. Στην κρίση των γαλακτοκομικών που προκλήθηκε από την κατάργηση των ποσοστώσεων. Και εγώ σας βεβαιώνω δεν θέλω να επανέλθουμε στο παλιό καθεστώς των ποσοστώσεων γιατί κάτι τέτοιο θα ήταν και στην σφαίρα του φαντασιακού. Είναι προφανές ότι δεν μπορεί να γίνει πλέον αυτό, αλλά οι ποσοστώσεις όπως ήταν διαμορφωμένες τότε βέβαια δεν ικανοποιούσαν όλους. Δεν μιλώ λοιπόν γι' αυτό, αλλά είδαμε στην κρίση των γαλακτοκομικών μετά από ένα χρόνο κρίσης, μετά από τεράστιες ζημίες σε βάρος των ε, παραγωγών, των αγροτησών και των αγροτών. Φανταστείτε τα σε νούμερα. παίρνουν τη Γερμανία, μόνο τα νούμερα για τη Γερμανία. 10 λεπτά αναλύτρο γάλακτος έχαναν. Έχαναν. Και μάλιστα μια χρονιά 15 σεντ. Μιλούμε για 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ που δεν κατέληξαν, δεν κατέληξαν στους Γερμανούς γαλακτοπαραγωγούς. Μεγάλη ζημιά για τους ε, παραγωγούς και για τη γερμανική υπεθρό. Τεράστια ζημία. Και μετά από ένα χρόνο εντατικότατε συζητήσεις στην Επιτροπή Γεωργίας μεταξύ των χωρών μελών. Επανήλθαμε στην κοινή οργάνωση αγοράς και καταλήξαμε σε ένα πρόγραμμα όπου οι γαλακτοπαραγωγοί που ε, μειώνουν εθελοντικά λαμβάνουν μια αποζημίωση. Και αυτό λειτουργήσε. Έχουμε και ένα παρατηρητήριο για το γάλα, το οποίο παρατηρεί τις κινήσεις της αγοράς. Και εάν εκεί εγκαταστήσουμε κάποιους μηχανισμούς που όταν θα δουν ότι μειώνεται η τιμή κατά ένα ποσοστό, χτυπάνε τα πρώτα καμπανάκια του κινδύνου. Και όποιο μειώνει του δίνεται ένα κίνητρο. Και όταν συνέλθει πια η αγορά μπορεί πάλι να απελευθερωθεί η παραγωγή. Γιατί να μην παράγει κανεί αν υπάρχει όντω αγορά για το προϊόν του, αλλά γιατί να παράγει όταν δεν υπάρχει αγορά, όταν απλώ συμπιέζεται η τιμή. Και μάλιστα εκείνη την εποχή είχαμε και τις υψηλότερε εξαγωγές. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι έμειναν στάσιμε οι εξαγωγές. Δηλαδή παρήγαμε για μια αγορά που δεν υπήρχε. Και ξαναλέω, έχουμε ακόμα 90.000 τόνους. Ίσως κάποιους από αυτούς να τους πουλήσαμε από τότε που κοίταξα τα νούμερα. Αλλά εξακολουθούν οι τόνοι αυτοί, 90.000 τόνοι, να συμπιέζουν τις τιμές στην αγορά. Δεν, δεν χρειάστηκε να δημιουργήσουμε νέους μηχανισμούς. Αν υπάρχει ένας μηχανισμός ώστε να μην χρειαζόμαστε κάθε φορά να περνάμε ένα ολόκληρο χρόνο συζητώντας πολιτικά, νομίζω τότε μπορούμε να προχωρήσουμε πολύ καλύτερα. Υπάρχουν συγκεκριμένες προ, προτάσεις, δεν μιλούμε για φαντασία. Όταν υπάρχει υπερπαραγωγή, έχουμε τους μηχανισμούς για να του προσαρμόζουμε, για να προσαρμόζουμε μάλλον την παραγωγή, στις ανάγκες αγορά. αγοράς. Αυτό μπορεί να γίνει και αυτοματοποιημένα. Όπως είπα, για το γάλα έχουμε ήδη παρατηρητήριο. Δεν είναι κάτι λοιπόν το οποίο, όπως είπα, καλούμεθα να επινοήσουμε στη βάση της φαντασίας, είναι κάτι το οποίο υπάρχει και μπορεί να εφαρμοστεί. Σας ευχαριστώ πολύ για τις προτάσεις που κάνατε ως τώρα. Αναμένω με μεγάλο ενδιαφέρον τις τροπολογίες και βεβαίως θα καταβάλω προσπάθεια να συνεργαστούμε επικοδομητικά, ώστε να μπορέσουμε να περιλάβουμε κάποια θεμελιώδη ενδιαφέροντα της ε, πολιτικής αναπτύξεως στην ε, υπόθεση αυτή της αναθεωρήσεως της ΚΑΠ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ Μαρία. Προθεσμία για τις τροπολογίες 5 Δεκεμβρίου 12 το μεσημέρι και η ψηφοφορία στην Επιτροπή θα γίνει στις 21 και 22 Ιανουαρίου του 2019. Αύριο το πρωί, 20 Νοεμβρίου, θα ξαναβρεθούμε για να ψηφίσουμε. 20 Νοεμβρίου είναι μια ημερομηνία πολύ σημαντική για οποιονδήποτε δημοκράτη στη χώρα μου την Ισπανία. Σας ευχαριστώ πολύ.